Good morning, colleagues. Um, a warm welcome to everyone. σας καλώς ήρθατε. Ιδιαίτερος καλώς ορίζω τους Ρουμάνους συναδέλφους και υπουργού τον κύριο Τουάντερ και την κυρία Ντανιέλα Ντάν. Πριν ξεκινήσουμε το πρώτο σημείο, το πρώτο ουσιαστικό σημείο της ε, παρουσίαση των προτεραιοτήτων τη Ρουμανική Προεδρία, να σα κάνω μερικέ ανακοινώσει. Καταρχήν, η οθέτηση ημερησία διάταξη. Έχουμε μερικέ αλλαγές. Σημείο 27. Ε, η έκθεση για την, το προσχέδιο συμφωνίας για, τη για την συνεργασία μεταξύ Eurojust και Γεωργία θα λάβει χώρα στι 10 και 30 αντί στις 11 και 40. Σημείο 26. Τροπολογίες για την δημιουργία του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας θα λάβει η χώρα συζήτηση στις 10 και 50 αντί για τις 11 και 20. Στις 1, 23 25 για τις θεωρήσεις θα λάβουν χώρα, θα συζητηθούν στις 11 και 10. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, να εγκρίνουμε την μερίσια διάταξη όπως τροποποιείται. Έγκριση πρακτικών της 27 Σεπτεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται. Γλωσσικό προφίλ συνεδρίαση. Έχουμε όλε τι γλώσσε εκτό από τα νέζικα, κροατικά και Ιρλανδικά και μερικές ε, ανακοινώσεις για κατεξοδότηση πράξης, δύο-τρεις συγκεκριμένα. Ε, μετά από αιτήματα πολιτικών ομάδων, εστάλησαν πολιτικέ κοινοποίησει στο Συμβούλιο των για, την, για, την, για τα αιτήματα παράταση προ ε, προθεσμιών ελέγχου για δύο θέματα. Ε, τον κανονισμό ε, τη 14-12-18 ε, που τροποποιεί το παράρτημα 2 του κανονισμού 5-15-14 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερική Ασφάλεια. Επίσης, ο κανονισμός του 14-12-18 που τροποποιεί το παράρτημα 2 του 516 του 2014. Στις 16 Ιανουαρίου 19 το Κοινοβούλιο έλαβε ε, τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, για την ανταλλαγή, συστηματική ανταλλαγή με ηλεκτρονικά μέσα ε, των πληροφοριών που σχετίζονται με πυρβόλα όπλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βασική πράξη είναι η Οδηγία 91-477 της 18 Ιουνίου 91 για τον έλεγχο και την κατοχή ε, και την απόκτηση όπλων. Ο συνήθως η πράξη αυτή κοινοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ε, μέσω του ΛΥΜΠΕΔΙΑ, ε, επιστολής 18 Ιανουαρίου 2019. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, παρακαλώ πολύ ενημερώστε τη γραμματεία για, μέχρι τις 30 Ιανουαρίου. Τέλος, 21 Ιανουαρίου 2019 η Κομισιόν κοινοποίησε την έναρξη διαβούλευση για μια πράξη κατεξιοδότηση για τι τρίτε χώρε ψηλού κινδύνου. Ε, θα ενημερωθούν και θα το, το θέμα θα συζητηθεί με την ομάδα εμπειρογνωμόνων για το ξέπλυμα χρήματο ε, και την τρομοκρατή, τη χρηματοδότηση ε, με γραπτή διαδικασία 23 από τις 23 Ιανουαρίου 2019, εφαρμοστικές πράξεις 10 Ιανουαρίου 2019, ε, απόφαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από την Ιαπωνία. Ε, βασικός κανονισμός, ο 216 ε, η λήψη αυτής της ε, πράξης κοινοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Αν έχετε κάποια αντίρρηση, ενημερώστε τη γραμματεία μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2019. Περνάμε στο πρώτο ουσιαστικό σημείο της ημερησίας διάταξης. Σας παρουσιάζω τους, ε, τους δύο υπουργού που έρχονται στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Οι εισηγητέ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι ήδη έχουν συναντηθεί με την Ρουμανική Προεδρία, οπότε έχουμε ήδη ξεκινήσει ε, αυτέ τι επαφέ και κάποιου τριμερεί διαλόγου. Χαίρομαι λοιπόν που η δουλειά έχει ήδη αρχίσει. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους Υπουργούς αλλά και όλα τα στελέχη της Ρουμανικής Προεδρίας. Καταρχήν λοιπόν να καλωσορίσω τον κύριο Τούντορελ Τοάντερ, Υπουργό Δικαιοσύνη και την κυρία Κάρμεν Ντανιέλα Ντάν, Υπουργό Εσωτερικών τη Ρουμανία. Χαίρομαι που είστε μαζί μα για να μα παρουσιάσετε τις προτεραιότητε τη Ρουμανική Προεδρία στα θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της δικαιοσύνη και των εσωτερικών υποθέσεων. Υπουργό, η κυρία Ντάν θα ξεκινήσει, αν καταλαβαίνω καλά, με τη δική τη ε, παρουσίαση. Ο, ο Υπουργό ε, Δικαιοσύνη ε, σα κατέστησε ε, εθελόντρια να ξεκινήσετε. Έχουμε συμφωνήσει οι παρουσιάσει σα να διαρκέσουν 10 με 12 λεπτά, κάθε μία. Κατόπιν θα ακολουθήσει συζήτηση θα δώσουμε το λόγο στους συντονιστές και τα μέλη για ερωτήσεις. Οι Υπουργοί ως συνήθως θα απαντήσουν ομαδοποιώντας ε, κατά θέμα τις ερωτήσεις. Αυτό που κάνουμε συνήθως δηλαδή. Ξεκινάμε λοιπόν με την Υπουργό, κυρία Ντάν, Υπουργό Εσωτερικών της Ρουμανίας. Παρακαλώ. Thank you very much, Mr. President. Κύριε Πρόεδρε Μωράης, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ ενώπιόν σας για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες αυτού του εξαμήνου όσον αφορά τις εσωτερικές υποθέσεις. 12 ε, χρόνια μετά την ένταξή μας, Θέλαμε και εμείς να συνεισφέρουμε για μια πιο συνεκτική Ευρώπη και πιο δυνατή. Η άσκηση της Προεδρίας είναι ύψης της σημασίας, είναι πολύ σοβαρό καθήκον και γνωρίζουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε περίπλοκα ζητήματα και για τους πολίτες και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις εσωτερικές και εξωτερικές όπως η απόσυρση της Μεγάλης Βρετανίας, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η πολιτική γειτονία που δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Γι' αυτό θα θέλαμε να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της περίοδου και αυτών των δράσεων και τι συνέπειες θα υπάρχουν για την Ένωση και την συνοχή της. Κάθε φορά που αναλύσαμε με τους συναδέλφους τα ζητήματα αυτά, τους φακέλους αυτούς, για να δούμε τι δράσεις πρέπει να αναλάβουμε για να προχωρήσουμε αυτά τα θέματα. Θέσαμε το εξής ερώτημα πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε εμείς στις ανησυχίες, τους φόβους και τις προσδοκίες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ακολουθήσουμε γοργά βήματα για ένα από τα θέματα που μας απασχολούν τις ευρωεκλογές. Και γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι καθήκον μας είναι να ακούσουμε τη φωνή των Ευρωπαίων πολιτών και να κατανοήσουμε τις προσδοκίες τους. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των μελημάτων και της προσοχής μας. Γι' αυτό οι αξίες της ευρωπαϊκής μας οικογένειας θα πρέπει να προωθηθούν. Αξιότιμα μέλη. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας δυσκολεύει είναι η μάχη που πρέπει να δώσουμε με το χρόνο. Γιατί θα πρέπει ο ρυθμός συζητήσεων να είναι πολύ εντατικός και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και διαθέσιμοι από το σύνηθες. Θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις στα τρία θεσμικά όργανα και μέσα σε μία ομάδα του Συμβουλίου για να βρούμε τα καλύτερα μέσα με γοργά βήματα. Θα, θέλουμε, θα θέλαμε και εμείς να προωθήσουμε τα ζητήματα που μας απασχολούν επικοδομητικά. Και νομίζω ότι συμμεριζόμαστε τους ίδιους στόχους. Μία Ευρώπη που ευημερεί, που είναι ενωμένη, που είναι συγκλητική και που πλησιάζει τους πολίτες της και φυσικά να είναι και ένας παγκόσμιος παράγοντας. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε θεμελιώδεις αρχές που μας διέπουν πάντα για την ασφάλεια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Κατά την άποψή μας αυτές οι αρχές ισχύουν και θα πρέπει να αποτελέσουν τον θεμέλιο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί πρόκληση αλλά και ευκαιρία. Υπάρχουν απειλές που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανένα κράτος από μόνο του. Και φυσικά υπάρχουν επιπτώσεις στους πολίτες πολλών κρατών. Υπ' αυτή την έννοια η συνοχή μεταξύ κρατών μελών αποτελεί βασικό πυλώνα ο οποίος θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή πέρα από τις ε, δηλώσεις προθέσεων. Υπό αυτό το πνεύμα θα κινηθούμε και θα λάβουμε υπόψη την ήδη προϋπάρχουσα ατζέντα. Υπ' αυτή την έννοια θα συνεισφέρουμε άμεσα στην ε, παγιοποίηση των θέσεών μας και γι' αυτό ζητώ την υποστήριξή σας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις προσπάθειες και τη συνεργασία σας. Κυρίες και κύριοι, η ε, ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας, η διαχείριση των εξωτερικών σύνορων καθώς και η διαχείριση του χώρου Σέγγεν, η πολιτική θεωρήσεων, η μετανάστευση και το προσφυγικό είναι ζητήματα ύψης της σημασίας. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τα βασικά ορόσημα που έχουμε κατά νου σε σχέση με την ε, παγιοποίηση της εσωτερικής ασφάλειας, όπως ξέρετε, η τρομοκρατική απειλή είναι ένα μείζον ζήτημα και γι' αυτό ακριβώς στις 11 Δεκεμβρίου 2018 είδαμε μία άλλη απειλή να φανερώνεται στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου. Γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία που δεν έχει σύνορα. Η Επιτροπή κατά της τρομοκρατίας ε, συνέταξε μία έκθεση και θα λάβουμε υπόψη τις συστάσεις σε επίπεδο Συμβουλίου για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, αναδίους, αναδιόμενη απειλή κατά της ασφάλειάς μας. Επίσης, στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Τζάι, ε, θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα και χαίρομαι διότι ο πρόεδρος σας, ο Κλοντ Μοράις, μας είπε ότι θα συμμετάσχει στις εργασίες. Κατά τη διάρκεια της Άνοιξης θα οργανώσουμε μία διάσκεψη, θα λάβετε προσκλήσεις φυσικά για την ε, καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές. Θα προβούμε σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για να αντιμετωπίσουμε επιγραμμικά και μη την ριζοσπαστικοποίηση και για να προστατεύσουμε τους πολίτες προβλέπεται συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρμοδίων αρχών. Κατά την άποψή μας θα πρέπει να ενισχύσουμε το προληπτικό σκέλος στα επόμενα χρόνια. Θεωρούμε σημαντική τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών σε αυτή την προσπάθεια καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης οι πολίτες στο κοινωνικό τους περιβάλλον μπορούν να δουν ορισμένες αλλαγές συμπεριφοράς που είναι εξωτερικά ε, δείγματα ρίζοσπαστικοποίησης σε συμπολίτες τους. Επίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλουμε να καταπολεμήσουμε αυτή την μάστιγα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εξεύρουμε τις ε, κατάλληλες λύσεις για την ε, πρόληψη και ε, διαχείριση των αιτίων αυτής της κακοδαιμονίας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τις πληροφορίες οικονομικών συναλλαγών των τρομοκρατών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις επιγραμμικές δραστηριότητες των ενδυνάμει τρομοκρατών. Ξέρω ότι έχετε πολύ φορτωμένη ατζέντα, αλλά θα θέλαμε να μην αφήσετε κατά μέρος, να μην αναβάλλετε αυτή την πρωτοβουλία. Γι' αυτό ακριβώς θα προωθήσουμε την πολιτική στα πλαίσια του 18 μέχρι το 22. Το Συμβούλιο προβλέπει μέτρα σε στρατηγικό επίπεδο αλλά και επιχειρησιακό για να προωθήσουμε την εσωτερική μας ασφάλεια. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τα ναρκωτικά, ε, έχουμε την δεκάτη επέτειο των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών. Στις 14 και 15 Μαΐου λοιπόν στη Βιέννη θα γίνει μία συνάντηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Η Προεδρία μας θα καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να καθοδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη σε αυτή τη διαδικασία διαπραγματεύσεων. Σε σχέση με την εξωτερική διάσταση της ασφάλειας, το 2018 κίνησε ένα πιλωτικό σχέδιο σε σχέση με ε, τους πυρήνες εγκλήματος υπό το, την ονομασία Σοφία. Ήδη από τον Νοέμβριο είχαμε πολλές πληροφορίες σε σχέση με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς συνεργασίας. Το Συμβούλιο υποστηρίζει αυτή την καινοτόμο πρωτοβουλία και το Μάρτιο του 19 θα ασχοληθούμε στο Συμβουλίο με το θέμα αυτό. Δηλαδή θα λάβουμε υπόψη την ε, τεχνολογία και την κινητικότητα για να λάβουμε υπόψη τις ε, πολυπολιτισμικές ιδιαιτερότητες που διαγράφονται στα κράτη-μέλη. Το ίδιο το μέλλον της Ευρώπης ε, βασίζεται στις δικές μας προτεραιότητες που μπορεί να διαφέρουν από κράτος σε κράτος. Όχι όμως κατά Θα θέλαμε να προωθήσουμε αυτές τις δράσεις με εντατικούς ρυθμούς για την ασφαλειά μας. Θα θέλαμε έναν ανοιχτό και επικοδομητικό διάλογο με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάλληλη υποστήριξη για τους στόχους μας σε σχέση με την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Έχει μεγάλη σημασία η διασφάλιση των εξωτερικών μας συνόρων και η διαχείριση του χώρου Σέγγεν. Θέλουμε να προωθήσουμε λύσεις για διαπραγματεύσεις, για την ε, ακτοφυλακή και την συνοριοφυλακή, έτσι ώστε να ενισχυθούν για την εξασφάλιση ασφαλέστερων συνόρων. Η ε, διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφορικής και πληροφοριών στον κυβερνοχώρο έχει μεγάλη σημασία. Η Προεδρία μας θα προωθήσει τις ε, διαπραγματεύσεις για έναν κανονισμό για τις ενιαίες ευρωπαϊκές ταυτότητες καθώς και τις άδειες διαμονής με βάση την αλλαγή του κώδικα Σέγγεν που θα εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με το μηχανισμό αξιολόγησης του χώρου Σέγγεν η Προεδρία θα επιταχύνει τη διαδικασία για τις ε, συστάσεις μέσα στα πλαίσια των αξιολογήσεων και σχεδίων δράσης στα κράτη-μέλη. Στον τομέα της μετανάστευσης, η Ρουμανική Προεδρία θα συνεχίσει τις συζητήσεις για την αναγνώριση και εξέβρεση λύσεων από τα κράτη-μέλη μέσα στα πλαίσια της σωστής ισορροπίας μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης για να γίνει πιο αποδοτικό το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με βάση τον κανονισμό χορήγησης ασύλου και τις προόδους που έχουν επιτελεστεί. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε ε, μία συμφωνία σε σχέση με τους συνδέσμους μεταξύ κρατών μελών. Ως προς την μείωση των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης είναι προτεραιότητα. Θα θέλαμε να υποστηρίξουμε την ΕΙΕΔ καθώς και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς για να έχουμε συνεργασία με τη χώρα προέλευσης και τις χώρες διαμετακόμισης. Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να μειώσουμε τους οικονομικούς και παράνομους μετανάστες. Σε σχέση με το καθεστώς θεωρήσεων, η Ρουμανική Προεδρία θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Θεωρήσεων και τον κανονισμό που σχετίζεται με την επικαιροποίηση στοιχείων ως προς τις θεωρήσεις. Θα προωθήσουμε και τις συζητήσεις σε σχέση με τα ενδεχόμενα μέτρα συνεχούς κατάρτισης των υπευθύνων σε σχέση με την κοινή πολιτική θεωρήσεων. Σε σχέση με την πολιτική προστασία, η Προεδρία θα προσδώσει μεγάλη σημασία στην πολιτική προστασία, ανθρωπιστική βοήθεια και διαχείριση κρίσεων. Στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σε σχέση με τον φανισμό πολιτικής προστασίας. Θα ε, λάβουμε υπόψη την διαδικασία προπαρασκευής από τα κράτη-μέλη και αυτό συλλογικά, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε καταστάσεις ε, κατεπίγουσας ανάγκης και απρόβλεπτα γεγονότα που θα μπορούσαν να έχουν κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς αντικτύπους. Κύριε Πρόεδρε Μωράης, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, αυτές ε, είναι οι βασικές αρχές και ορόσημα που θα ήθελα να σας κοινοποιήσω στην αρχή της συνάντησής μας Περιμένω τις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών στη συνέχεια. Τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τουντορέλ Τόουντερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, για δεύτερη φορά βρίσκομαι ενώπιον σας και αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα. Για να σας παρουσιάσω συνοπτικά τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας και για να προσπαθήσω να απαντήσω στις ε, τυχόν ερωτήσεις σας. Ως Υπουργός Δικαιοσύνης θα ήθελα καταρχήν να τονίσω ότι εκτιμώ προσωπικά πάρα πολύ το έργο σας και το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί μέσω της νομοθεσίας που προωθείτε εκπροσωπείτε την δημοκρατική νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αυστριακή Προεδρία με την οποία συνεργάστηκα στενά στο παρελθόν διότι διευκόλυνε την προετοιμασία μας και την προώθηση των φακέλων και ζητημάτων που μας απασχολούν, καθώς και ορισμένες πρωτοβουλίες που αρχικά προώθησε η Αυστριακή Προεδρία. Θα θέλαμε να έχουμε στενή συνεργασία μαζί σας με την Επιτροπή, αλλά και προσωπικά και μεμονωμένα με ευρωβουλευτές, αν το επιθυμούν, γιατί έτσι μόνο θα φτάσουμε στους στρατηγικούς στόχους που ορίζονται μέσα στα πλαίσια του νομοθετικού μας ε, μελήματος. Σίγουρα θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που προβλέπετε. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε συνένεση εκεί που είναι δυνατόν και όπως προείπα θα φτάσουμε στους συμβιβασμούς εκεί που γίνεται γνωρίζω το τεράστιο έργο σας καθώς και το έργο των προηγούμενων προεδριών στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων έτσι ώστε να προωθήσουμε πολιτικές υπέρ των πολιτών και να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της δικαιοσύνης, καθώς και την εμπιστοσύνη των πολιτών για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί περίοδος προκλήσεων, αλλά είμαι πεπισμένος ότι θα τις ε, αντιπαρέλθουμε και θα φτάσουμε στους ε, επιθυμητούς στόχους κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής ε, Προεδρίας ή δυνατόν. Θέλουμε η Προεδρία να είναι αποτελεσματική και να βασίζεται στην ε, στενή μας συνεργασία. Μια Προεδρία που να στρέφεται προς αποτελέσματα, απτά αποτελέσματα δεν θα πτωηθούμε καθόλου. Θα προωθήσουμε τις κοινέ μας αξίες καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου, σεβόμενοι τις ε, ε, παραδόσεις και τα διάφορα δικαιοδοτικά συστήματα των κρατών μελών μέσα στα πλαίσια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης των συστημάτων δικαιοδοσίας στα κράτη-μέλη. Θα σας κάνω κι εγώ μία παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας στον τομέα της δικαιοσύνης και αυτό θα το κάνω συνοπτικά έτσι ώστε να μην χάσουμε χρόνο α, για τις ερωτήσεις σας. Γι' αυτό θα σας μιλήσω για τα θέματα τα οποία έχουμε ήδη ενώπιόν μας και που απασχολούν και την Επιτροπή σας. Υπ' αυτή την έννοια θα αναφερθώ στην ανάγκη έγκρισης κανονισμού για τα ηλεκτρονικά στοιχεία και τις ηλεκτρονικές αποδείξεις στον τομέα του ποινικού δικαίου, την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία σε περιπτώσεις ποινικού. Εγώ ως ε, επικεφαλής ε, του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θεωρώ ύψης της σημασίας αυτό το ζήτημα, διότι τη στιγμή που υπάρχει διασυνοριακή εγκληματικότητα, η οποία ολοένα και αυξάνεται και επειδή Έχουμε και συνεργασία των δικαστικών αρχών. Γνωρίζουμε τις τελεσίδικες αποφάσεις των κρατών μελών και γι' αυτό χρειάζεται στενή συνεργασία και στην αρχή της διαδικασίας καθώς και στην ε, παρακολούθηση της πορείας της. Έχουμε λοιπόν αυτό τον κανονισμό και την σχετική οδηγία χρειάζεται εξισορρόπηση ως προς την πρόληψη της εγκληματικότητας και την αντιμετώπιση της για λόγους δημοσίας τάξης. Και φυσικά θα πρέπει να σεβαστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ατομική προστασία του πολίτη. Μας ενδιαφέρει το δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον και όπως ε, έχει αποφανθεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας ενδιαφέρουν θέματα δημόσιας τάξης χωρίς να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των κρατών μελών μέσα στα πλαίσια των ε, ε, δικαιωμάτων και ελευθεριών. Με τη δική σας ε, συμμετοχή θα βρούμε αυτή την σωστή ισορροπία. Το, το Δεκέμβριο το ε, Συμβούλιο Υπουργών ΖΑΗ ασχολήθηκε με αυτό το σχέδιο κανονισμού και θα συνεχίσουμε αυτή τη, με αυτή μας την προσέγγιση και για το σχέδιο οδηγίας. Το ταχύτερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη το γενικό συμφέρον, αλλά και την αποφασιστικότητά μας να αποδώσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ζίπελ, την εισηγήτρια, γιατί πέρσι συζητήσαμε αυτά τα θέματα. Είχαμε μία πολύ καλή συνεργασία έτσι ώστε το Συμβούλιο να κάνει τα κατάλληλα βήματα το ταχύτερο δυνατόν για την ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου και ιδιαίτερα της οδηγίας. Επίσης υπάρχει ένα άλλο συναφές ζήτημα. Η θέση σε εφαρμογή παγιοποιημένης συνεργασίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ χρειάζεται ε, μία επιχειρησιακή δραστηριότητα η οποία είναι απολύτως απαραίτητη. διότι ε, ήδη υπάρχουν τρεις-τέσσερις ε, δικαστές που πλαισιώνουν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εισαγγελίας για να προστατεύσουμε τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εγκληματικότητα δεν έχει σύνορα. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε τα μέσα καταπολέμησης αυτού του φαινομένου διευρωπαϊκά και διεθνώς. Μίλησα για ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία να πρέπει να, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε σε εφαρμογή αυτόν τον κανονισμό, έτσι ώστε όπως ξέρετε στο εγγύς μέλλον θα διοριστεί ο επικεφαλής εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Αρχής καθώς και το Διευθυντήριο. Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία η οποία έχει κινήσει και το Νοέμβριο 2020 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο της ε, καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Η Ρουμανική Προεδρία θα προωθήσει τις συζητήσεις διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας η οποία εκδηλώνεται διαφορετικά ανάλογα με το που εκδηλώνεται και φυσικά υπάρχει και το φαινόμενο νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων. Ένα άλλο ε, θέμα αφορά τις, ε, το θέμα της παραχάραξης των χρημάτων. Μπορέσαμε να φτάσουμε σε μία συμφωνία για την υποβολή της οδηγίας κατά την Αυστριακή Προεδρία και γι' αυτό χρειάζεται ε, αγαστή συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ρουμανική Προεδρία θα ήθελε να συνεχίσει τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο για την ολοκλήρωση της οδηγίας αυτής. Και όταν δοθεί τελική μορφή στο κείμενο από την νομική υπηρεσία, και εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, θα το εντάξει η Προεδρία στην ατζέντα του Συμβουλίου για την τελική έγκριση. Επίσης, προσδίδουμε μεγάλη σημασία στο πρόγραμμα αξιών, αξιών της δικαιοσύνης διότι πέρα από το αστικό, ποινικό ή εμπορικό δίκαιο, σημασία έχουν οι κοινέ μας αξίες και άκρο σημαντική είναι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών για τον εκδημοκρατισμό της. Και η Ρουμανική Προεδρία θα καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να έχουμε μία γενική ενωσιακή προσέγγιση. Φυσικά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που εκκρεμούν, όπως ο κανονισμός για την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων ως προς το οικογενειακό δίκαιο, δαιμονία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα θέματα αποτελούν προτεραιότητα. Θα ήθελα να κάνω και μια μικρή παρένθεση. Αυτές οι κανονιστικές πράξεις έχουν ήδη αρχίσει να ε, τίθενται σε εφαρμογή. Ακολουθούμε επιταχυμένους ρυθμούς και πιστεύω ότι ως από κοινού νομοθέτες θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτό το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο έτσι ώστε να ε, ολοκληρώσουμε το καθήκον αυτό, το οποίο μας τιμά ιδιαίτερα. Μέσα στα πλαίσια της Προεδρίας βεβαίως θα μπορούσα να παρουσιάσω και άλλα ζητήματα, θα το κάνω το απόγευμα όμως στα πλαίσια των εργασιών άλλης επιτροπής. Ξέρω ότι έχω υπερβεί το χρόνο μου, σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ και αναμένω τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. thank Ευχαριστώ πολύ και τους δύο υπουργούς Και προχωρούμε τώρα στις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Όλοι οι συναδελφοί βεβαίως θέλουν να μιλήσουν. Είναι ανοιχτά όλα τα θέματα ε, τώρα στο τέλος της ε, θητείας μας, σημαντικά θέματα. Και γι' αυτό λοιπόν, για να προλάβουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις, θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να περιοριστούν στα δύο λεπτά ομιλίας. Και μετά μπορούμε να δώσουμε ένα δεύτερο γύρο αν χρειαστεί. Ρομπέρτα Μετσόλα, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί Υπουργοί, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα και εύχομαι καλή επιτυχία για την πρώτη αυτή Προεδρία. Σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαστε καλοί και υποστηρικτικοί εταίροι. η ομάδα μου. Πιστεύει ότι η, η Ρουμανία έχει θέση στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Προεδρία της θα πρέπει να αποτελέσει υπόδειγμα ευρωπαϊκών αξιών και για την Ένωση αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Γι' αυτό και παραλαμβάνω, κυρίες, κυρία και κύριε Υπουργέ το, τη δήλωση και τη θέση ότι η διαφθορά είναι ακριβώς στους αντίποδες των ευρωπαϊκών αξιών. Γι' αυτό μας ανησυχούν τα προβλήματα που βλέπουμε στη Ρουμανία. Πρέπει να τα καταπολεμήσουμε με κάθε τρόπο. Ιδάλλως θα αρχίσει να παρουσιάζει ροχμές στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και όχι μόνο στη δική σας χώρα, ούτε στη δική μου μόνο, αλλά σε όλη την Ένωση. Οι Ρουμάνοι πολίτες βλέπουμε να υψώνουν την ευρωπαϊκή σημαία παρά το πολικό ψύχος. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε και να καταστέλλονται οι ειρηνικές διαδηλώσεις από τη ρουμανική ε, κυβέρνηση. Ε, είναι λοιπόν οι ειρηνικοί διαδηλωτές, είναι φιλοευρωπαίοι, φιλοευρωπαίοι ε, ακρεφνείς οι Ρουμάνοι και είμαι βέβαιη ότι δεν πρόκειται να τους, να τους εγκαταλείψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο και το λέμε αυτό γιατί βλέπουμε ότι χιλιάδες κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν τους τελευταίους μήνες. Εσείς επιμένετε πως τα α, γεγονότα αυτά, οι αποφυλακίες δηλαδή οφείλονται στον συνοστισμό στις φυλακές. Θεωρείτε λοιπόν ότι πρέπει να κατασκευαστούν νέα κτίρια σοφρενιστικών ιδρυμάτων, ή να ε, διευρυνθούν οι εγκαταστάσεις των υφισταμένων ή πρέπει να αποφυλακίζονται οι κρατούμενοι. Και επίσης μπορείτε να δεσμευτείτε πως δεν θα προχωρήσετε σε περαιτέρω ε, τροποποιήσεις ή να θεωρήσεις τις ε, ε, νομοθεσίας για τη δικαστική εξουσία χωρίς να ε, λάβετε υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Τι μέτρα θα λάβετε προκειμένου να μην επαναληφθούν τα γεγονότα που είδαμε πρόσφατα και επίσης τι σκοπεύετε να κάνετε για να διευκολύνετε τον διάλογο για την ακτοφυλακή για να κλείσει πριν από τις ευρωεκλογέ του Μαΐου. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, συνάδελφοι, όμως να μην ξεπερνάτε τα δύο λεπτά γιατί δεν πρόκειται να αφήσουμε αρκετό χρόνο για τους λοιπούς συναδελφούς. Η κυρία Σίπλη, εκ μέρους των Σοσιαλιστών Δημοκρατών, σήμερα είναι ασθενής, αλλά νομίζω ότι ο Γιώ, Λάινεν, ο Γιώ να Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Με σύντομο χρονικό διάστημα, βέβαια, στη διάθεσή η Ρουμανική Προεδρία θα έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής και έχοντας ακούσει με μεγάλη χαρά τις ε, δεσμεύσεις για, τα, για την αλληλεγγύη. Θα ήθελα βέβαια να ξέρω τι σημαίνει αυτό και για το πακέτο του ασύλου που έχει κατατεθεί από το Κοινοβούλιο. Είστε διατεθειμένοι να το προωθήσετε γιατί εμείς βλέπουμε με απογοήτευση οι βουλευτές ότι το Συμβούλιο δεν κάνει δεκτές τις δικές μας ε, παρενέσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να ρωτήσω και επίσης για την μπλε κάρτα όπου βλέπουμε πως δεν υπάρχει καμία πρόοδος ενώ θα έπρεπε ε, να βρούμε κάποιες λύσεις που θα συνδυάζουν αυτή την ε, νέα διαδικασία με την πολιτική της μετανάστευσης γιατί παρα, ε, παραπέμπεται στα, σκα, στα σκαλένδα αυτή την πρόταση για την μπλε κάρτα εργασίας για τους μετανάστες. Ε, επίσης, εσείς έχετε το τελευταίο διάστημα της βουλευτικής περίοδου, της βουλευτικής αιτίας. βλέπετε ότι θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε θέματα που έχουν μεγάλη σημασία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, γιατί υπάρχει βέβαια ο κανονισμός για την, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά όχι για τον ιδιωτικό βίο. Δηλαδή έχουμε το GDPR, αλλά έχει το privacy. Ε, μπορείτε να προωθήσετε λοιπόν και το privacy εγκαίρως πριν από το τέλος της ε, περίοδου. Η Ρουμανία, ξέρουμε, θα έχει πάρα πολλή δουλειά να ολοκληρώσει. και οπωσδήποτε θα χρειαστεί να συνεργαστείτε για να με την Επιτροπή για να εξασφαλίσετε και με τις κοινοβουλευτικέ επιτροπές του Κοινοβουλίου για να εξασφαλίσετε πρόοδους. Ε, οι διαδικασίε ε, του άρθρου 7 κατά της Πολωνίας και της Ουγγαρίας επίσης πέφτουν στο δικό σας εξάμεινο. Έχετε εσεί υπόψη κάποια περαιτέρω βήματα για το Κοινοβούλιο. Ήταν μεγάλη απογοήτευση που δεν υπήρξε πρόοδο στι ε, διαδικασίε κατά τη ε, Ουγγαρία, τουλάχιστον στου προηγούμενου μήνε. Ευχαριστώ πολύ, Χέλγα Στίβεν. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Καταρχήν να ξεκινήσω με την κατάσταση όπως υφίσταται αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία. Η Ρουμανία είναι ένα σημαντικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νεότερο από τα Παρ' παρόλα αυτά είναι το κράτος το οποίο δημιουργεί τις περισσότερες ανησυχίες. Λαμβάνοντα υπόψη το κράτος δικαίου και την κατάστασή του στη Ρουμανία, την ε, ανεξαρτησία του δικαστικού, της δικαστικής εξουσίας, ε, εξετάσαμε προσεκτικά το ψήφισμα που υιοθετήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Ελπίζω και εσείς να το διαβάσατε καλά και σας ζητούμε να αποφύγετε την υιοθέτηση οποιονδήποτε μέτρων που θα νομιμοποιούσαν στην πράξη τη διαφθορά. Η, η πιο πρόσφατη έκθεση για την ε, Ρουμανία ήταν και η πιο ανησυχητική. Θα θέλαμε λοιπόν να μας απαντήσετε σε αυτές τις επικρίσεις ε, τις οποίες περιλαμβάνει. Το σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της Ρουμανικής Προεδρίας. Ευχαριστούμε την, ε, για την παρουσίαση του προγραμματός σας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα εξής εκ μέρους της ομάδας μου. Η Ειδική Επιτροπή για την κατά της τρομοκρατίας. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα θέλαμε ε, να ε, προχωρήσουμε στο θέμα της απόσυρσης ε, τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο. Ελπίζουμε ότι εκεί θα προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό και χαιρόμαστε που το έχετε και εσείς ως προτεραιότητα. Μια άλλη δική μας προτεραιότητα είναι η διαλειτουργικότητα Μια βάση δεδομένων, ευρωπαϊκή βάση δεδομένων βιομετρικών στοιχείων στο διαδίκτυο, ηλεκτρονική δηλαδή, θα ήταν πολύ σημαντική και θα βελτίωνε την αποτελεσματικότητα των δράσεών μας για την εσωτερική ασφάλεια. Χαιρόμαστε που και αυτό είναι μεταξύ των δικών σας προτεραιοτήτων. Έχουμε και άλλα πολλά σημαντικά θέματα να σχολιάσω απλώς το θέμα του, της μεταρρύθμισης του ασύλου και της μετανάστευσης. Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσέγγιση πακέτου και να ψηφίσουμε ένα-ένα τα θέματα χωριστά. Για παράδειγμα, το σύστημα Eurodac για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ε, η, ε, η συνάδελφος ε, από τα δεξιά μου, κάθε δεξιά μου, ε, έχει υποβάλει μια πολύ καλή πρόταση και θα θέλαμε να προχωρήσουμε, να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτήν. Δυστυχώ πρέπει να... Υπάρχει κάποια πρόοδος στο θέμα αυτό της μεταρρύθμισης του ασύλου και της μετανάστευσης. Ευχαριστούμε. Κυρία Κρίσμπεκ θα ήταν εδώ, αλλά το, λόγο για αυτήν θα πάρει η κυρία Ιντφελτ για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστούμε πολύ για, τα, για την παρουσίαση του προγράμματος της Ρουμανικής Προεδρίας. Θα ήθελα και εγώ, όπως και οι προηγούμενες δύο μιλήτρες, να εκφράσω την βαθιά μου ανησυχία για το κράτος δικαίου και την κατάστασή του στην Ρωμανία και για τη διαφθορά, για, την, για θέματα ε, συνεργασίας μεταξύ δικαστικού και αστυνομικού σώματος. Ε, το ευρωπαϊκό σύστημα θα λειτουργήσει και σε αυτό το επίπεδο και σε επίπεδο ευρωπαϊκής ε, εισαγγελίας μόνο αν όλα τα κράτη-μέλη σέβονται τις ίδιες προδιαγραφές ε, και τους ίδιους κανόνες. Οπότε η εσωτερική σας πολιτική θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές σας φιλοδοξίες και με ανησυχία μαθαίνουμε ε, τα περί της ε, ενδεχόμενης ε, αναστολής, ακύρωσης μάλλον, ε, καμιάς, ε, περίπου μιας εκατοσταριάς δικαστικών αποφάσεων καταδίκης για θέματα δωροδοκίας και διαφθοράς. Η κυβέρνησή σας θα πρέπει να εφαρμόσει τι ε, συστάσει Επιτροπή Βενετία σε ό,τι αφορά τι νομοθετικέ αλλαγέ που χρειάζονται. Για το πακέτο του ασύλου, άκουσα τον Υπουργό να λέει ότι θα αναζητήσετε ευρεία ε, συμπαράσταση, ευρεία ε, υποστήριξη. Δεν χρειάζεστε ευρεία υποστήριξη, χρειάζεστε απλή πλειοψηφία. Αυτό λέει η συνθήκη. Το Συμβούλιο λοιπόν να πάρει απόφαση και να τελειώνουμε. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε μέχρι να εξασφαλίσετε ομοφωνία. Δεν χρειάζεστε ομοφωνία. Οπότε σας ενθαρρύνουμε να κλείσετε αυτό το πακέτο κατά διάρκεια της Προεδρίας σας. Επίσης, αναφερθήκα στο πρόγραμμα δικαιωμάτων και αρχών. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι σκοπεύετε να ολοκληρώσετε τη συζήτηση και υιοθέτηση αυτού του πακέτου κατά διάρκεια της Προεδρίας σας. Τέλος, αν μιλάμε για αρχές, τι προσκοπεί να κάνει η Ρουμανική Προεδρία για να αναζωογονήσει την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων που βαλτώνει εδώ και περίπου 10 χρόνια. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, αν εξακολουθήσετε να υπερβαίνετε το χρόνο που σας έχει δοθεί, θα έχουμε πρόβλημα αργότερα. Δύο λεπτά για τον καθένα, αυστηρά παρακαλώ. Η FTD και το ENF δεν έχουν αντικαταστάτες, οπότε θα μιλήσουν αργότερα. Παρακαλώ πολύ, όχι πάνω από δύο λεπτά όμω έτσι. Προχωράμε. Ο κ. Κουέλιο. Α, ζητώ συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Πριν από εσά, κύριε Κοέλιο, έχουμε του πράσινου. Κύριε Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Προεδρία θα πρέπει να δίνει το παράδειγμα. Πάντοτε. Πρέπει να αποτελεί παράδειγμα και υπόδειγμα για του υπόλοιπου. Το γεγονό ότι η Ρουμανική Προεδρία ε, δέχθηκε ε, μετανάστες από, τις, ε, από τα, τα, πλεούμενα αυτά πριν από δύο εβδομάδες ήταν πολύ καλό από το Sea-Watch. Ε, θα πάρετε μια παρόμοια πρωτοβουλία και στο μέλλον με το Sea-Watch. που θα μπορέσουμε να καταλήξουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική που δεν θα χρειάζεται κάθε φορά να διαπραγματευόμαστε, κάθε φορά δηλαδή που σώνονται κάποιοι άνθρωποι στη θάλασσα να διαπραγματευόμαστε μεταξύ μα για το ποιο θα του δεχτεί. Πάμε παρακάτω. Τώρα, η πρωτοβουλία του κ. Τόντερ για την ε, ακύρωση εκατοντάδων καταδικών ε, για διαφθορά δεν νομίζω ότι είναι καλό παράδειγμα. Επίσης μιλάτε για την αμοιβαία εμπιστοσύνη ως ε, βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς την υποσκάπτετε, διότι υποσκάπτετε την δικαστική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο, ή πρωθυπουργό σα, ε, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, μίλησε για τέσσερις πυλώνες. Ένας από τους πυλώνες της Προεδρίας σας, υποτίθεται θα είναι οι Ευρωπαϊκές Αρχές. Πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Δεν το βλέπω όμως ακόμα. Εγώ ως εισηγήτρια για τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 της συνθήκης για την Ουγγαρία ζήτησα συνέντευξη και ε, συζήτησα να βρεθούμε, να συναντηθούμε και το αρνηθήκατε. Πώς σκοπεύει το Συμβούλιο να ε, προσεγγίσει τις διαδικασίες του άρθρου 7 για την Ουγγαρία και την Πολωνία. Ε, τι έχει πει ως τώρα το Συμβούλιο. Το, η προηγούμενη Προεδρία μάλλον είπε ότι όλα αυτά επαφίονται στην επόμενη Προεδρία, τη Ρουμανική. Ε, εσείς πώς σκοπεύετε να, τι συνέχεια σκοπεύετε να δώσετε. Δώστε το παράδειγμα. Αυτό περιμένουμε από εσά. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά, ένα δευτερόλεπτο. Κύριο Κοέλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ του δύο υπουργού. Δύο ερωτήσει. Πρώτη, η είσοδο τη Ρουμανίας και Βουλγαρία στη ζώνη Ζέγγεν. Ήμουν εισηγητή το 2011. Το Κοινοβούλιο είναι συνεπές σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα στις εκθέσεις τους. Και στην τελευταία έκθεση του κ. Στάνισλεφ ε, επιμείναμε σε αυτή την ιδέα. Δεν θέλουμε οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι πολίτες να εξαιρεθούν του ζώνη Σέγγεν. Ερώτηση. Η Προεδρική Ρουμανία θα υποφεληθεί τη προεδρία τη προκειμένου το θέμα αυτό να μπει στην ημερησία διάταξη και να λήξει. Δεύτερη ερώτηση. Δεν είναι πολύ διαφορετική από αυτή που έθιξαν άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχουν πολλέ ανησυχίε σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα. Ενοχλεί που το, το, θέμα του ασύλου στο Συμβούλιο έχει μπλοκαριστεί τελείω. Ε, πέντε κράτη-μέλη έχουν ελέγχους στα σύνορά τους. Αυτό παρεμποδίζει την κυκλοφορία των προσώπων. Και έχουμε και το σύστημα VIS, ε, στο οποίο τίθενται θέμα, θέματα ορισμού, ορισμών. Οπότε η ερώτηση είναι, εξαιτία των ε, ευρωεκλογών έχουμε λίγο χρόνο. Ποια είναι τα νομοθετικά κείμενα, τα νομοθετικά θέματα, ντοσιέ, στα οποία θα εστιάσετε. Δεν είναι δυνατόν να ε, μοιράσουμε τις δυνάμεις μας σε πολλά ζητήματα. Οπότε ποιες είναι οι πολιτικές, προεδρίες, οι πολιτικές προτεραιότητες της Προεδρίας ποια από, τα, ποιοι από τους νομοθετικούς φακέλους ε, που βρίσκονται αυτή στην τραπέζι σας πιστεύετε ότι μπορούν να συζητηθούν και να κλείσουν σε αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα που έχουμε. Ο Απρίλιος είναι η τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν τις εκλογές. Ποια θέματα πιστεύω θα μπορούσαν να κλείσουν μέχρι τότε. Thank you very much, Mr. Mrs. please. Η κυρία Μακουβέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ο πληθυσμός της Ρουμανίας αξίζει του σεβασμού όλων. Έγιναν πολλές διαμαρτυρίες στους δρόμους, πολλές διαδηλώσεις στη Ρουμανία. Όλοι θέλουμε μία πολύ καλή Ρουμανική Προεδρία. Αλλά θα πρέπει να σας πιστεύουν τα κράτη-μέλη όταν είσαστε επικεφαλής, όταν είσαστε επικεφαλής της Ο κύριος Κατάινεν είπε ότι χρειάζεται σεβασμός όταν, και γιατί το είπε ο κύριος Κατάινεν, όταν χτες το ακυρωτικό δικαστήριο μοίρασε συγχωροχάρτια στην κυβέρνηση και χτες η Πρωθυπουργό είπε ότι μίλησε με σας κύριε Υπουργέ Τόντερ έτσι ώστε αυτά τα διατάγματα να περάσουν το συντομότερο ε, και να ισχύσουν έτσι ώστε να δοθεί άφεση στη διαφθορά. Για να είσαστε επικεφαλής ε, του Συμβουλίου ΖΑΗ και για να αποτελέσετε παράδειγμα, αυτό που έχει σημασία είναι ακριβώς τι κάνετε. Σε σχέση με αυτή τη συγκαλυμμένη αμνηστία την αναλαμβάνετε, δεν είσαστε υπόλογοι για αυτήν. Ξέρετε ότι η Ρουμανία μπορεί να δεχτεί κυρώσεις για αυτά τα μέτρα αμνηστίας. Αναφέρεται επίσης στις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας ότι θα υποστηρίξετε και την επέκταση τα δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά της ε, τρομοκρατίας. Έχετε υπερβεί τα δύο λεπτά. Όχι, όχι, όχι, τελευταία πρόταση. Ε, όλοι πρέπει να αρκεστούν στα δύο λεπτά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ε, ισχύει για την καταπολέμηση της απάτης. τι θέλουμε να κάνουμε, να ξεπεράσουμε αυτό το ζήτημα της απάτης και να σταθούμε σε κάτι άλλο, κύριος Πάβελ. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας, αλλά και για τις ε, προτεραιότητες που δείχνουν ότι είμαστε αρκετά φιλόδοξοι. Δεν έχω ερωτήσεις γιατί μελέτησα το πρόγραμμα. Ζήτησα το λόγο για να σας, ε, ε, για να, ε, για να σας πω τι είπε η προλαλή να σταθώ σε αυτό. Ε, σας μίλησε μία πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης που ενέκρινε τον ποιητικό κώδικα ε, χωρίς δημόσια συζήτηση. Αυτός ο ποινικό κώδικας που εγκρίθηκε από την πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης ε, θεωρήθηκε από το ακυρωτικό δικαστήριο ένας άκυρος νόμος ε, και αυτό αφορά το συνταγματικό δίκαιο, το σύνταγμά μας που εγκρίθηκε το 2003 πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης υπενθυμίζει τι έγινε. Εγώ ως νέος ε, και επειδή ε, δεν έζησα την επανάσταση θα ήθελα να αναλύσετε και την θέση της κυβέρνησης σε σχέση με, την ε, επίγουσα, με το επίγον διάταγμα. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ποιος μιλάει πριν κρίνουμε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Έχετε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο και σας συγχαίρω γι' αυτό. Η Σιλβίκη Γιώμ. Ε, θα προσπαθήσω να συνεχίσω κι εγώ. Να πάρω τη σκητάλη είπε και η κυρία Σαρχεντίνη για τους πυλώνες και τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Και θα ήθελα συμμεριζόμενος και τα ανησυχίες των συναδέλφων να αναφερθώ σε ένα ζήτημα. Τη νομοθετική πρωτοβουλία για το η κοινωνική πτυχή, τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, τον αγώνα κατά των διακρίσεων για λόγους φύλου. Και θα ήθελα κύριε Πρόεδρε, ε, και έχω τόσο λίγο χρόνο να πω, τι έχετε να πείτε για την ε, Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης και την κύρωσή της. Ευχαριστώ, Ντάλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους υπουργούς που ήρθαν εδώ για την ε, παρουσίαση αυτή. Σας εύχομαι βεβαίως κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Σας ευχαριστώ που μας επισημάνατε τις, τις προτεραιότητές σας. Η διαχείριση της ε, η βιώσιμη διαχείριση και αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης ε, με απασχολεί εμένα. Μιλήσατε για καλές λύσεις, συνενετικές λύσεις. Αυτό σημαίνει για μένα ότι θα επιδιώξετε συνένεση της κάθε πλευράς. Πώς θα το καταφέρετε αυτό. Βλέπουμε τεράστιες αποκλήσεις στο θέμα της μετανάστευσης, ενώ ορισμένοι δεν θέλουν καν να μοιραστούν το βάρος. Και μιλάτε για ιδιαίτερες δυνατότητες των κρατών μελών. Πώς θα το διαχειριστείτε αυτό, το θέμα των διαφορετικών δυνατοτήτων των κρατών μελών. Εμεί τώρα έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το διάστημα τη μια κρίση πάνω στην άλλη. Μακροχρόνιες λύσεις δεν έχουμε, μόνο ad hoc λύσεις υιοθετούμε, οι οποίες, και αναφέρομαι εδώ συγκεκριμένα στη Μάλτα, κράτος πολύ μικρό, επομένως λοιπόν χωρίς μακροπρόθεσμες λύσεις πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ισορροπημένη αντιμετώπιση. Και μια και δεν έχω χρόνο μεταρρύθμιση λέτε στο σύστημα, στο κοινό σύστημα ασύλου. Η συγγήτρια είμαι εγώ για το Ταμείο Μετανάστευσης και Ασύλου και θα ήθελα να ξέρω τι είδους χρονοδιάγραμμα έχετε υπόψη για το θέμα του ασύλου και για το Ταμείο βεβαίως. Κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργή για την συνοπτική παρουσίαση της ατζέντα σας. Θα ήθελα να πω ότι έχετε τέσσερις μήνες αντί για έξι στη διάθεσή σας και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους που μίλησαν επί του θέματος και όχι για την κατάσταση στη Ρουμανία. Διαφορετικά θα έπρεπε και ε, εμείς να σταθούμε σε άλλα ζητήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κοέλιο που ε, τόνισε ότι θα έπρεπε ε, να ενταχθούν στο χώρο Σέγγεν μετά από το 2011 που κάναμε την αρχική αίτηση, μετά από 16 προεδρίες. Θα πρέπει να ληφθεί μία απόφαση επί του θέματος. Την επόμενη εβδομάδα στην Μίλνη Ολομέλεια έχουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση, την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης. Γιατί αυτό αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς θα αντιμετωπίσετε έμπρακτα τη ριζοσπαστικοποίηση. Ως μέλος της Επιτροπής της Βενετίας θα ήθελα ε, να σας ρωτήσω πώς ορίζεται το κράτος δικαίου, γιατί υπάρχουν και αιρεσιμότητες εκτός συνθήκες και αν θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, νόμος για να είναι υπόλογη οι δικαστές, οι δικαστικές αρχές. Ο κύριος Σόγκορ και εγώ θα μιλήσω στα ρωμανικά. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανοιχτά ζητήματα και τα οποία θα πρέπει να ολοκληρηθούν. Θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία. Οι συνάδελφοι Κοέλιο και Γκραπίνη υπενθύμησαν το θέμα του Σέγγεν. Πώς θα μπορέσετε να προωθήσετε το θέμα. Τώρα θα συνεχίσω στα Ουγγρικά. Και θα ήθελα να αναφερθώ στα προβλήματα αυτά που αναφέρθηκαν, διαφθορά, κράτος δικαίου, αλλά θα σταθώ στις διακρίσεις. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχετε μπορέσει να αντιμετωπίσετε στο εσωτερικό της χώρας σας. Γι' αυτό λοιπόν δεν γίνεται δεκτό η, η της Επιτροπής ε, σε σχέση με το θέμα της ουγγρικής μειονότητας. Γιατί δεν γίνεται δεκτή η σημαία στην περιοχή αυτή, τα σύμβολα δηλαδή. Ευχαριστώ κύριος Νίτερ Μιούλερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ναι και δεν έχω τόσο χρόνο, θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Προς την Προεδρία η ερώτηση είναι τι συγκεκριμένα βήματα σκοπεύετε να αναλάβετε προκειμένου να σημειωθούν βήματα στις προτάσεις για τη μετανάστευση και το άσυλο. Φρόντεξε παραδείγματι, γιατί έπονται ψηφοφορίες, ε, ΕΑΖΟ. Ήδη υπήρξε συμφωνία το 2017 για το, με το Συμβούλιο για το θέμα της ΕΑΖΟ, αλλά πρόοδος δεν έχει σημειωθεί έκτοτε. Άλλη ερώτηση. Καθώς δεν βλέπω καμία πιθανότητα να εξασφαλιστεί πρόοδος ε, για, το, για τη συμφωνία του Δουβλίνου, για την αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου, η Ρουμανική Προεδρία διαβλέπει κάποια πιθανότητα για προσωρινή έστω συμφωνία αναδιανομής όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διασχίζουν τη Μεσόγειο και δεν γίνονται δεκτοί σε κανένα λιμάνι ευρωπαϊκής χώρας, βλέπετε εσείς η Ρουμανική Προεδρία τη δυνατότητα να ε, γίνουν δεκτοί με σύστημα αναδιανομής με όποια κράτη θέλουν ε, εθελοντικά να συμμετάσχουν ε, και να τους υποδεχθούν. Δηλαδή να δώσουμε μια λύση έστω ανθρωπιστικής φύσεως προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γιούρεκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στη Ρουμανία κατά τη ε, ε, διάρκεια της Προεδρίας της, να επιτύχει περισσότερη συνεργασία, αλληλεγγύη, σεβασμό, αλληλοκατανόηση κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πως η συνεργασία στηρίζεται σε συνθήκες και σε όχι, όχι σε αυθαίρετες αποφάσεις. Άρα πρέπει να διευθετούνται οι διαφορές και οι συγκρούσεις με βάση τους νόμους, τους κανόνες και όχι με τρόπο αυθαίρετο. Έτσι λοιπόν το αίτημα για αποκλεισμό της της Πολωνίας ε, από την ε, διαδικασία λήψη αποφάσεων του Συμβουλίου ε, απερίφθη, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία 4 πέμπτων, έχει κλείσει δηλαδή το θέμα. Και ναι, μπορεί κανείς να θέλει να τροποποιεί τις συνθήκες, αλλά δεν μπορεί να τις παραγνωρίζει. Και για τη Ρουμανία. Πρέπει να πει το Συμβούλιο ξεκάθαρα ότι η ψηφοφορία της 12 η Σεπτεμβρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως έτοιμα για ε, εκκίνηση διαδικασίας του άρθρου 7. Γιατί δεν επετεύχθη η ε, πλειοψηφία του άρθρου 354. Εδώ είχαμε να κάνουμε με μια χονδροειδή κομμωδία. Πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες. Καμία σχέση δεν έχουν αυτά με τη δημοκρατία. Να κλείσουν αυτές οι υποθέσεις λοιπόν, να μειωθούν και οι εντάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμβάλλει και η Ρουμανία με τον τρόπο αυτό στην ε, ανανέωση του ε, σεβασμού του οποίου χαίρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Κινίτση, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ε, κυρία και τον κύριο Υπουργό για την παρουσία σου τους εδώ. Συγκεκριμένε ερωτήσεις λοιπόν. Ζητώ συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Προς τον Υπουργό των Εσωτερικών. Ε, αναφερθήκατε στη ριζοσπαστικοποίηση και την πρόληψη αυτής είτε διαγραμμικά, είτε εκτός, είτε στα σοφρονιστικά εδρήματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κύριε Υπουργέ, η πρόληψη της ρουσπαστικοποίησης δεν θα έπρεπε να περάσει και σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή μέτρων κοινωνικών και κυρίως παιδαγωγικού χαρακτήρα που θα δημιουργούσαν όρους συγκεκριμένης και απτής ε, ενσωμάτωσης κοινωνίας, γιατί είδαμε στη τελευταία τρομοκρατική επίθεση του Στρασβούργου, ε, ότι αυτή ε, την διέπραξε Ευρωπαίος πολίτης που είχε απλώς άλλο καταβολές. Επίσης, η διαχείριση του, της Τρομοκρατία τρομοκρατίας και τη μετώπιση της, που ξέρουμε ότι έχει αναπτύξει δίκτυα με ε, διακήρυξη ναρκωτικών ανθρώπων και πολλά ε, άλλες δραστηριότητες που εν τέλει χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Θα ήθελα να ρωτήσω και δεδομένων ε, και των πολλών συστάσεων της αρμόδιας ειδική επιτροπής για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Πώς σκοπεύετε και ξέρουμε βέβαια ότι είναι πολύ περιορισμένο το χρονικό διάστημα που έχετε θέσει σας να δώσετε κάποια περαιτέρω όθεση στις ε, προτάσεις αυτές και επίσης για τη συνεργασία την αστυνομική στην ανταλλαγή πληροφοριών που, έχει, που έχουν τεράστια σημασία για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών οργανώσεων και όχι μόνο της ε, τρομοκρατίας βέβαια αλλά όλων των εγκληματικών οργανώσεων. Τι είδους πρωτοβουλία σκοπεύετε να εισαγάγετε για την ε, προαγωγή συγκεκριμένων μέσων ε, που θα έχουν να κάνουν παραδείγματι με την ταυτοποίηση δραστών ποινικών ε, εγκλημάτων και κυρίως πάγωμα οικονομικών στοιχείων, περιουσιακών στοιχείων και επίσης για τις οικονομικές συναλλαγές, φόρος για τις, στοιχεία για τις οικονομικές συναλλαγές. Πώς μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τζεκόφσκι. Θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω πως η συζήτηση εδώ δεν πρέπει να αφορά, δεν αφορά τις, ε, τα εσωτερικά πολιτικά τεκτενόμενα της ε, Ρουμανίας και με ξαφνιά στο γεγονός ότι ορισμένοι εδώ ε, βρήκατε ευκαιρία να επιτεθείτε κατά των συναδέλφων σας. Έχετε υπόψη τι σημαίνει gentleman, τι σημαίνει αυρότητα, σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αξιοποιείτε την συνεδρίασή μας εδώ για να βάλετε κατά των συναδέλφων σας. Και δεύτερον, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Χαίρομαι που θα έχετε την ευκαιρία με την Προεδρία σας να αποδείξετε πως είστε μια χώρα σύγχρονη, μια χώρα ισχυρή, πως θέλετε να αλλάξουν κάποια πράγματα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Πώς αξιολογείτε τον ε, σύνδεσμο μεταξύ της, πρόσβαση, της πρότασης για την ε, επαναπροώθηση των παρανόμως διαμενόντων ε, αλλοδαπών και τη ΣΥΚΑ, το πακέτο δηλαδή για το άσυλο. Είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί ένα αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ για την συγκεκριμένη απάντηση που περιμένω να ακούσω. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριο Σκέστα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και θα αναφερθώ πρώτα στην ανθρωπιστική κρίση στη Μεσόγειο 2.200 παιδιά μεσήλικες, γυναίκες ε, ανήλικοι γυναίκες έχασαν τη ζωή τους ε, στην ε, Μεσόγειο προσπαθώντας να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν μπορεί η Ευρώπη να προτείνει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως ζητούν άλλωστε και οι οργανώσεις ε, βοήθειας προς τους ετούντες. Είστε διατεθειμένοι λοιπόν όταν ε, έχουμε οργανώσεις εθελοντών που κάνουν διάσωση από βέβαιο πνιγμό αυτών των ανθρώπων, μια λύση που θα επέτρεπε αυτόματα αυτοί οι άνθρωποι που κινδυνεύουν από πνιγμό να αναδιανέμονται στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις εβδομάδες χρειάστηκε να περάσουν, στην περίοδο μάλιστα μεταξύ Χριστουγέννων και νέου έτους λίγο πολύ, άνθρωποι πάνω σε ένα πλοίο ε, χωρίς κατεύθυνση να περιμένουν ποιο κράτος θα τους υποδεχθεί μέχρι να δοθεί μια λύση. Και για το άσυλο, μια Ευρώπη της αλληλεγγύης σημαίνει ταυτόχρονα την ανάληψη της ευθύνης όχι μόνο από το κράτος της πρώτης άφηξης όπως η Ισπανία, η Μάλτα, η Ιταλία. Αλλά εν τέλει αυτό το οποίο έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλληλέγγυα αναδιανομή των προσφύγων για να σταματήσει αυτή η αδικία της κατανομής των προσφύγων με βάση το, σύστημα του, το ισχύον σύστημα του ε, Δουβλίνου. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα τεράστιο επιτεύγμα της Ρουμανικής Προεδρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι ίσως θα ήταν σκόπιμο να πείτε δύο λόγια για τα βήματα που σκοπεύετε να αναλάβετε σε σχέση με την αντιμετώπιση της ε, κρίσης αυτής. Κυρία Σουάνα. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δραστηριότητά σας, την ε, επερχόμενη δραστηριότητά σας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία να θα ήθελα να μην σας κάνει εντύπωση ε, η δραστηριότητα ορισμένων ε, συναδέλφων μας, γιατί αν και είναι Ρουμάνοι, στην ουσία σπηλώνουν την ίδια τη Ρουμανία. Οι πληροφορίες υπάρχουν, ξέρουμε πως ε, έχουν. Η κυρία Μακοβέη που ελπίζω να μη συμμετάσχει σε κανένα από τα θεσμικά όργανα στο μέλλον, ήταν υπουργό Δικαιοσύνης και κατέστρεψε το δικαιοδοτικό σύστημα στη Ρουμανία. Εν μία νύχτη ε, άλλαξε όλους τους εισαγγελείς χωρίς ε, καμία δικαιοδοσία. Άλλαξε τον ποινικό κώδικα χωρίς ε, δημόσιες ε, διαβουλεύσεις και χωρίς να περάσει από το Κοινοβούλιο η πρόταση νόμου. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι αυτό. Την ερώτησή σας σας παρακαλώ λέει ο Πρόεδρος. Και εγώ επειδή είμαι νέα δεν μπορώ να δεχτώ μία τέτοια συμπεριφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έπρεπε να αναφερθώ σε αυτήν. Θα ήθελα να σας πω ότι η Ρουμανική Προεδρία θα είναι μία προεδρία προκλήσεων. Έχετε το Brexit, την ασφάλεια, το Frontex, ε, τη, τα εξωτερικά μας σύνορα τις προκλήσεις ασφάλειας και ούτω καθεξής. Ποιες είναι οι προοπτικές της Ρουμανικής Προεδρίας σε σχέση με τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, δεν γίνεται. Πρέπει να σταματήσετε. Τι θα γίνει με την ακτοφυλακή και τη συνοριοφυλακή. Έχετε υπερφεί κατά πολύ το χρόνο σας. Έχουμε μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μας κύριε Υπουργή. Δύσκολα θα απαντήσετε σε κάθε μία από τις ερωτήσεις χωριστά. 10 λεπτά ο καθένας πρέπει να ομαδοποιήσετε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, ζητήσω ο καθένας ε, να απαντήσει σε ερωτήσεις που τον αφορούν και σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του και δεύτερον ε, προσπαθήστε να ομαδοποιήσετε για παράδειγμα εισαγγελία, πακέτο ασύλου, οι συγητές είναι εδώ, το, το θέμα της σήμανσης του Βλήνου, τα σημαντικά θέματα, παρακαλώ πολύ να εστιάσετε σε αυτά, γιατί έχουμε περιορισμό χρόνου. Ε, οποιασδήποτε ερωτήσεις δεν μπορείτε να, δεν προλάβετε να απαντήσετε, μπορείτε να τις απαντήσετε γραπτός. Και αν υπάρχουν παράπονα λέω των ευρωβουλευτών, παρακαλώ πολύ να απευθυνθούν σε μένα και εγώ θα αναλάβω. Παρακαλώ τους υπουργούς να εστιάσουν στο τι μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια αυτής της Προεδρίας. μέχρι τον Απρίλιο βασικά στους δύο τομείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Ποιος θα ξεκινήσει? Η κυρία Ντάν. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές για τις ερωτήσεις που υπέβαλαν. Θα προσπαθήσω να τις διατρέξω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μετσόλα για τις εκτιμήσεις της. Σας ευχαριστώ και για τις ανησυχίες που εκφράσατε. Εγώ ασχολούμαι με την ασφάλεια των συνόρων, των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλώντας για τις πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ε, πέρυσι είχαμε λιγότερη πίεση. Η κορύφωση της πίεσης είχε γίνει το 2015. Αυτό σημαίνει ότι η απάντηση των κρατών μελών ήταν επαρκής επί το πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα λειτουργούν καλώς. Γνωρίζουμε απόλυτα αυτό το ζήτημα θα πρέπει να προβλέψουμε λύσεις και θα πρέπει να αντλήσουμε από τα διδάγματα του παρελθόντος. Εμείς θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε ώστε οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ε, σαφείς ε, και μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή θα πρέπει να εγκριθούν τάχιστα. Τώρα, σε σχέση με τη Frontex, με τον οργανισμό αυτό, θα ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες, ιδιαίτερα με τις χώρες των Βαλκανίων, για να αντιμετωπίσουμε το νομικό και νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση και με τις επιτόπιες ε, δράσεις και ομάδες. Αυτή η πρόταση υπάρχει από το Σεπτέμβριο πέρσι και μιλήσαμε και για απόσπαση εργαζομένων από άλλες χώρες, χώρες άμεσης γειτονίας. Νομίζω ότι ο διάλογος αυτός με τις τρίτες χώρες θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις και με άλλες χώρες. Ο κύριος Βάιντεν Χόισερ υπέβαλε μία ερώτηση. Ε, θα ήθελα να απαντήσω και στην κυρία Ελγα Στίβενς παράλληλα. Μου μιλήσατε για το Ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης ασύλου. Ε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρόκειται για ένα ε, άκρος σημαντικό χαρτοφυλάκιο και έχουν καταβληθεί σοβαρές προσπάθειες ε, για να γίνει πρόοδος και να βρούμε λύσεις. Ως προεδρεύουσα του ΖΑΙ θα ήθελα να σας πω ότι θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για την εξέβρεση λύσεων, θετικών λύσεων που να αντικατοπτρίζουν την εξισορρόπηση μεταξύ, την ισορροπία μεταξύ ευθυνών και αλληλεγγύης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Πολλοί μίλησαν για την ε, ΚΕΠΑ γενικότερα και ζητήματα τα οποία μπορούμε να δούμε και χωριστά. Θα θέλαμε τουλάχιστον να ε, ξεμπλοκάρουμε ε, μία συνιστός αυτού του πακέτου. Δεν υπάρχει απόλυτη σαφήνεια υπό αυτή την έννοια όσο και να θέλουμε να προχωρήσουμε και να δώσουμε τελική μορφή σε ορισμένα ε, νομοθετικά μέτρα σε σχέση με τον κανονισμό του Δουβλίνου έχουμε εντολή διαπραγμάτευσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Γνωρίζουμε τη σημασία εξέβρεσης λύσεων για την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου και για τη σωστή χορήγηση ασύλου. Θα μπορούσα να σας μιλήσω και για τη Eurodac και διάφορες επιμέρους οδηγίες. Θα ήθελα να σα εγγυηθώ ότι θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε σχέση με την πρόταση για τον κανονισμό για τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου συνεχίζουν οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Υποβάλλατε και μία ερώτηση και για τη μπλε κάρτα. Είμαι πεπισμένη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο γνωρίζει πώς έχουν οι διαθεσμικές διαπραγματεύσεις για αυτή τη διαδικασία της ε, μπλε κάρτας. Υπήρξαν πολλά προσκόμματα. Και οι θέσει των δύο θεσμικών οργάνων αποκλίνουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις προγενέστερες προεδρίες γιατί προσπάθησαν να προωθήσουν συγκεκριμένα πακέτα για την εξέβρεση ενός συμβιβασμού. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι καμία προσπάθεια δεν στέφθηκε από επιτυχία μέχρι τώρα. Φυσικά και η μετανάστευση έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα η παράνομη μετανάστευση. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την οδηγία της μπλε κάρτας για να βρούμε μία λύση που να μπορεί να είναι αποδεκτή και από, τους δύο, και από τις δύο νομοθετικές αρχές. Βεβαίως, εξαρτόμαστε από την υποστήριξη των κρατών μελών. Η κυρία Στίβενς μίλησε για την έκθεση που υποβλήθηκε για τη Ρουμανία και θα ήθελα να μιλήσω και από τη δική μου πλευρά Όσον αφορά τη δική μου αρμοδιότητα, γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθόρα και να ισχύσει το κράτος ε, δικαίου στην πληρότητά του. Θα ήθελα να κάνω και ένα άλλο σχόλιο, γιατί έχω ασχοληθεί και με την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς ως Υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων. Ε, ασχολούμαστε συνέχεια με την βελτίωση του γενικού πλαισίου και την καταπολέμηση καθώς και την πρόληψη της διαφθοράς. Ευχαριστώ και την κυρία Σαρτζεντίνη για το ερώτημά της. Μιλήσατε για το θέμα των μεταναστευτικών ροών και της κρίσης στη Μεσόγειο. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και δείξαμε την αλληλεγγύη μας ως προς αυτή την μεταναστευτική πίεση που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Για να ξεπεράσουμε αυτά τα γεγονότα, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μία συντονισμένη απάντηση από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε συνεκτικές δράσεις. Καθότι κατέχουμε την Προεδρία, ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να καταδείξουν την αλληλεγγύη τους και ε, εκτιμώ τη συνεισφορά των κρατών μελών που συνεισέφεραν άμεσα. Η χώρα μας και εκείνη με βάση το κανονισμό ε, του Δουβλίνου η χώρα μας δέχτηκε μετανάστες. Και στις 4 Δεκεμβρίου του 18 στο Συμβούλιο για την διαχείριση της μετανάστευσης θεωρήσαμε ότι μπορούμε να βρούμε και προσωρινές λύσεις για επιμέρους ζητήματα μέσα στα πλαίσια της άμεσης απάντησης ε, καταστάσεων κατεπίγουσας ανάγκης. Αυτό το είπαμε και στην Κορεπέρ και κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα αναλύσουμε το θέμα περαιτέρω και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Κύριε Κοέλιο, σας ευχαριστώ για τη θέση σας σε σχέση με την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στο χώρο του Σέγγεν και η συνθήκη του Άμστερνταμ κάνει μνήα στο κοινοτικό κεκτημένο και γι' αυτό θα έπρεπε να προσχωρήσουμε και εμείς να τεθεί σε εφαρμογή, δηλαδή το νομοθετικό πλαίσιο στο σύνολό του, δηλαδή να μην υπάρχουν έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα, κάτι που αντικατοπτρίζει τη Ρουμανία. Θεωρώ ότι στόχος προσχώρησης στο χώρο Σέγγεν ήταν στόχος μετά το 2007 θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεχή σας υποστήριξη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που στο σύνολό του εκφράστηκε υπέρ της προσχώρησής μας σε πολλές περιστάσεις. Και αυτό καταδεικνύει την αθέμητη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Οι πρόσφατες συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δείχνουν την ανάγκη λήψης απόφασης από το Συμβούλιο το ταχύτερο δυνατόν σε σχέση με τη θέση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Πληρούμε τους όρους ήδη από το 2011 και θα πρέπει να εφαρμοστεί το κεκτημένο του Σέγγεν. Φυσικά χρειάζεται μία προσέγγιση ενότητας επί του θέματος και να μην προβάλλουν προσκόμματα ορισμένα κράτη-μέλη. Όλοι όσοι έχουν επιφυλάξεις θα πρέπει να κατανοήσουν αυτή την επιχειρηματολογία. Η Ρουμανία δεν προτίθεται να υφίσταται ελέγχου, συνεχείς ελέγχου σε σχέση με το κοινοτικό και εκτιμένο τη στιγμή που πληρούμε όλους τους όρους, το έχουμε προβάλει πολλές φορές, έχουμε επιχειρηματολογήσει υπέρ αυτής της προσέγγισης και ελπίζω να βρισκόμαστε στην τελική φάση αποδοχής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τις ερωτήσεις επί του θέματος. Ο κύριος Ντεκόφσκι υπέβαλε ένα ερώτημα σε σχέση με το, το θέμα της οδηγίας για την επαναπρόθεση. Ίσως θα μπορούσα να επεκταθώ κάπως, αν και είπα ότι αυτό το θέμα είναι ύψης της σημασίας η επαναπροώθηση των πολιτών που βρίσκονται παράνομα στο ευρωπαϊκό έδαφος αποτελεί ένα βασικό πυλώνα της πολιτικής μετανάστευσης και νομίζω ότι είναι απόλυτα αναγκαίο να ε, δοθούν οι κατάλληλοι πόροι για όσους χρήζουν ε, γενικής προστασίας θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί σε σχέση με τον επαναπατρισμό και την επαναπροώθηση και θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την οδηγία περί επαναπατρισμού. Θα θέλαμε να γίνει πρόοδος, να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις το ταχύτερο δυνατόν. Βεβαίως το θέμα αυτό της ε, εσωτερικής ασφάλειας μπορεί να αποτελέσει και πρόκριμα για την εξέβρεση μιας συνολικής λύσης. Για να δούμε ποια είναι και τα εμπόδια για να προωθηθούν οι διαπραγματεύσεις. Θα μπορούσα να συνεχίσω επί μακρόν, αλλά θα πρέπει να αφήσω και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να απαντήσει. Θα ήθελα να σας ε, να, ε, να ευχαριστήσω και την ε, κυρία Μακοβέη. Θα ήθελα να μου είχε θέσει το ερώτημα για τη Eurodac, αλλά οπωσδήποτε θα προωθηθεί και αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι θα ήθελε βέβαια να σχολιάσετε και άλλα από τα ερωτήματα, αλλά ίσω θα ήταν σκόπιμο να δώσετε γραπτό απαντήσει απαντήσεις στις ερωτήσεις που δεν βρήκαν απάντηση στη συνεδρίες. Θα τις περιμένουμε συνάδελφοι, μια ο χρόνο ήταν αρκετά περιπιαστικό. Ο κύριο Υπουργό. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Θα ήθελα ότι, ελπίζω να μην κάνω λάθος τα ονόματα, η κυρία Μετσόλα είπε ότι η θέση της Ρουμανίας ε, είναι και θα πρέπει να είναι εντός χώρου Σέγγεν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην καρδιά μας και ελπίζουμε αυτό να ισχύει και αμφίδρομα. γιατί ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κοινό χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας, ελευθεριών και ασφάλειας, στον οποίο πιστεύουμε απόλυτα. Εγώ έχω καταγράψει όλες τις ερωτήσεις. Αν πρέπει να κάνω μία πρώτη μεγάλη ομαδοποίηση θα έλεγα ότι μου απευθύνονται ως προευρεύοντα του Συμβουλίου και άλλες ως ε, Υπουργού Δικαιοσύνης, ως Υπουργό Δικαιοσύνης. Θα προσπαθήσω εντάχει να απαντήσω. Εν πάση περιπτώσει θα απαντήσω στις περισσότερες ερωτήσεις. Κυρία Μακοβέη. Είπατε ότι θέλουμε να επεκτείνουμε να επεκτείνουμε τη δράση της Ευρωπαϊκής ε, Εισαγγελίας πριν ε, ε λειτουργεί. Όχι γιατί αυτό θα σήμαινε αλλαγή του άρθρου 86 των συνθήκων. Θα πρέπει να εξετάσουμε την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα συμπεράσματά του καθώς και τις προτάσεις της Επιτροπής. Μιλούσα για το μέλλον, δηλαδή μετά από την αρχή δραστηριοποίησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής. Διαφορετικά δεν θα ε, γινόταν κάτι τέτοιο δυνάμει του άρθρου 86 των συνθήκων. Ε, κράτος δικαίου. Αυτό που έχει σημασία να γνωρίζουμε ότι το κράτος δικαίου ακολουθεί διάφορες φάσεις σε διάφορα κράτη. Δεν ευθυγραμμιζόμαστε όλοι γιατί έχουμε διαφορετικά δικαιοδοτικά συστήματα και διαφορετική ιστορία ως προς το κράτος δικαίου και την ε, παγιοποίησή του. Το κράτος δικαίου θα πρέπει να λειτουργεί με βάση τις συνθήκες. Πολύ σωστό. Το κράτος δικαίου θα πρέπει να ενσωματώνει τα προστάγματα των συνθήκων. Το κράτος δικαίου είναι μία αναπόδραστη πορεία προς την οικοδόμηση και θα πρέπει να γνωρίσουμε αυτή την αναπόδραστη πορεία του προς την οικοδόμηση και την παγιοποίηση με βάση τις ε, κωδικοποιημένες συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, ε, συστάσεις που δεν είναι κοινέ για όλους γιατί το κράτος δικαίου έχει διαφορετικό τρόπο οικοδόμησης και στάδια από ένα κράτος μέλος στο άλλο. Διαφορετικά θα υπήρχαν ε, εναρμονισμένες συστάσεις προς όλους. Θα πρέπει να τονίσουμε αυτά τα προαπαιτούμενα που ισχύουν διαφορετικά από, κράτος μέλος, από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο. Και φυσικά τα ανώτερα ε, δικαστήρια, τα ακυρωτικά δικαστήρια ακολουθούν ε, μια συγκεκριμένη πορεία, όπως είδαμε και στην περίπτωση της Πολωνίας. Θα πρέπει να ε, θεωρήσουμε ως πρόκριμα λοιπόν το νομοθετικό έργο Κάνατε ένα σχόλιο στο οποίο συμφωνώ. Θέλουμε να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και να αυξήσουμε τα πρότυπα ορθότητας. Δεν έχει νόημα κανένας να σπηλώνει τη χώρα προέλευσης του. Εγώ εργάζομαι αυτή τη στιγμή για έναν κοινό ποινικό κώδικα, δηλαδή έχω μελετήσει τον ποινικό κώδικα των περισσότερων κρατών μελών και σε αυτή την περίπτωση ξέρω ότι όταν λιδωρείται ένας εκπρόσωπος του κράτους υπάρχουν κυρώσεις. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με ένα άλλο ζήτημα στο οποίο δεν θέλω να επεκταθώ. Σε σχέση με το πρόγραμμα αρχών και αξιών θα προχωρήσουμε και επειδή πρέπει να σας απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι, θα ολοκληρώσουμε το κανονιστικό πλαίσιο εκεί όπου μπορούμε. Πιστεύω ότι αναφερθήκατε επιμακρών σε επιμέρους ζητήματα και ως προς τους κινδύνους του συστήματος δικαιοδοσίας στη Ρουμανία και του κράτους δικαίου. Και μιλήσατε για το κατεπήγον διάταγμα για την ακύρωση 100 ε, καταδικών περίπου. Θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να βασιστούμε πάντα στις σωστές πληροφορίες σε σχέση με την έκδοση αυτών των διαταγμάτων. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε τις ε, πληροφορίες ως προς αυτά τα συμφραζόμενα. Νομίζω ότι ε, οποιαδήποτε εθνική απόφαση τηρεί τα δικαιοδοτικά δεδομένα και αυτό αφορά και το δικό μας ακυρωτικό δικαστήριο. Δηλαδή, από το 2014 έχει αναθεωρηθεί το δικαιοδοτικό μας σύστημα. Και από το 2014 και μετά ε, αποσύρθηκαν δικαστές τη στιγμή που υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία καταπάτησης του δικαίου. Το συνταγματικό δικαστήριο ακολούθησε αυτή την πορεία μετά το 2014 και Το συνταγματικό δικαστήριό μας αποφάνθηκε ότι ορισμένοι εισαγγελείς έκλεισαν πρωτόκολλα και ανέθεσαν καθήκοντα διαφορετικά από αυτά που προβλέπονταν σε, σε περίπτωση ποινική δίωξης. Κανένας δεν θέλουμε να ε, μην τηρήσει αυτό το πλαίσιο. Όλοι θα τιμωρηθούν εκεί που πρέπει. Το συνταγματικό δίκαιο και το συνταγματικό δικαστήριο ορίζει να ξανανοίξουν αυτά τα πρωτόκολλα και στην περίπτωση καταδίκης και στην περίπτωση ακύρωσης της απόφασης γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την καταδίκη. Γι' αυτό ανοίγουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Αυτό δεν αφορά μόνο τις καταδίκες, αλλά όλες τις υποθέσεις κατά το χρονικό αυτό διάστημα στο οποίο προαναφέρθηκα. Πώς τηρούμε τις αποφάσεις και συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Τη σεβόμαστε με βάση το συνταγματικό μας πλαίσιο. Η Επιτροπή της Βενετίας είπε μην ε, ανακαλέσετε τα μέλη του ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου. Μην ανακαλέσετε αυτά τα διατάγματα σε περίπτωση που υπάρχει δίωξη. Και γι' αυτό εμείς κάναμε τις ανάλογες αλλαγές δικαστές μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σύμφωνα με τον νόμο μετά από 20 χρόνια επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Η σύσταση της Επιτροπής Βενετίας ε, ανέφερε ότι δεν πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο. Και έτσι οι ε, δικαστικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά από 20 χρόνια υπηρεσίας, διότι έχουμε 7.500 δικαστικούς που υπάρχονται σε αυτή την κατηγορία και θα είχαμε ένα ε, έλλειμμα δικαστών αν γινόταν κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις και ανησυχίες που εκφράστηκαν προσπάθησα να τις ομαδοποιήσω, αλλά σε άλλες ε, δεν απάντησα. Και γι' αυτό θα κάνω αυτό που πρότεινε ο πρόεδρος. Θα υποβάλω τις απαντήσεις μου γραπτώς. Σας ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, συνάδελφοι, αν νομίζετε ότι υπάρχουν ερωτήσει που δεν απαντήθηκαν, πέστε μου το και θα ζητήσω από τους υπουργούς να σας απαντήσουν γραπτός. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να μην απαντηθούν οι ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κουέλιο, έχετε κάτι διαδικαστικό. Μάλιστα, πρόεδρε. Είπατε ότι ζητήσατε από τους υπουργούς να απαντήσουν γραπτώς αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να απαντήσουν προφορικά. Ε, τέθη από πολλούς συναδέλφους ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που έχει σχέση με τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας σε ό,τι αφορά τα νομοθε... τους νομοθετικούς φακέλους. Στην... Η τελευταία ολομέλεια του Κοινοβουλίου είναι του Απριλίου στο Στρασβούργο. Το Συμβούλιο αποφάσισε να μην ξεκινήσει καινούριου τριμερείς διαλόγου μετά το Φεβρουάριο. Οπότε είναι σημαντικό η Επιτροπή, οι Υπουργοί να μας απαντήσουν ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Ποια, ποιοι νομοθετικοί φάκελοι, ποιους νομοθετικούς φακέλους σκοπεύετε να κλείσετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Αυτό <laughs> δεν ήταν διαδικαστικό ζήτημα, προφανώς. Κύριε Κοέλιο, ξέρω, είστε σας εκτιμώ πολύ. Δεν φαντάζομαι ότι σπαθήσατε να ε, αποφύγετε την εφαρμή του κανονισμού μας. Ε, η Προεδρία μας ανέφερε, γιατί οι εκπρόσωποι της Προεδρίας μας ανέφεραν ποιες θα είναι οι προτεραιότητές τους. Ε, η κατάσταση είναι πιεστική λόγω χρόνου, είναι μια διαδικασία που εξ, εκτιλήσεται αυτή τη στιγμή. Αν τους ε, ζητήσω να απαντήσουν, ρητά δεν νομίζω ότι θα μας ε, ε τι μπορούν να τελειώσουν μέχρι το Φλεβάρι είναι δύσκολο να το πούν. Έχουμε τόσους πολλούς φακέλους με πολύ μεγάλο αριθμό ανοιχτών θεμάτων. Οπότε ε, η δέσμευση υπάρχει, αλλά πρακτικά τι θα τελειώσει είναι δύσκολο να το πούμε. Συζήτησα και πριν με τους υπουργούς και γνωρίζουν το θέμα αυτό. Θέλετε παρόλα αυτά να πείτε κάτι για, αυτό, αυτήν την ερώτηση και ζητώ συγγνώμη στους συναδέλφους ε, που είναι υπεύθυνοι για τα επόμενα θέματα και είναι εδώ, εδώ και ώρα και περιμένουν. Θέλετε να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση ξανά μήπω για τις νομοθετικές σας προτεραιότητες. Θα μπορούσατε να πείτε μια-δυο φρασούλες και να τελειώσουμε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, λέει κυρία Ντάν. Δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση που δεν είναι. Νομίζω όμως ότι από την παρουσίασή μας κατέστησε σαφές ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε όλους τους φακέλους. Θεωρούμε ότι όλοι οι φάκελοι είναι σημαντικοί και θέλουμε να ολοκληρωθούν, να κλείσουν. Είναι δύσκολο να σας πω πόσους φακέλους θα κλείσουμε ή πόσους θέλουμε να κλείσουμε. Δεν εργαζόμαστε απομονωμένοι, συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο. Είναι δύσκολο να προκαταβάλουμε τι θα κάνουν οι υπόλοιποι φορείς, τα υπόλοιπα όργανα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε όλα τα μέτωπα. Να σας Υπενθυμίσω επίσης αυτό που είπαμε και αυτό που είπε και η Πρωθυπουργό μας παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες μα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ρουμανική Προεδρία εστιάζεται με ρεαλισμό και φιλοδοξία στα θέματα που θα αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας πρόθεσή μας είναι να σημειώσουμε πρόοδο στους τριμμένους διαλόγους. Και επιθυμία μας είναι να κλείσουμε το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό θεμάτων. Ορισμένες, ε, ορισμένοι φάκελοι, ορισμένα θέματα είναι πιο ίσα από κάποια άλλα, ε, για να παραφράσω τον George Orwell, Ε, αντίθετα με τα όσα είπε ο πρόεδρος Κομισιόν, ε, η, προεδρία, η Προεδρία είναι οργανωμένη, είναι αποτελεσματική και έχει αποφασιστικότητα. Τώρα, φίξατε θέματα όπως το πακέτο και το Δουβλίνο. Ε, αυτά είναι θέματα με τα οποία θα χρειαστεί, τα οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν. Τι θα γίνει με αυτά, τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι προτεραιότητες, αλλά είναι και στο περιθώριο της οικονομίας ε, τα πιο πολλά από τα θέματα. Όλα αυτά όμως είναι προτεραιότητες. Οπότε οι εισηγητές ε, είναι προσιλωμένοι, το κοινοβούλιο σε ψηλό επίπεδο είναι προσιλωμένο στο έργο αυτό. Οπότε η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ε, ότι το με, η μεγάλη ερώτηση του Κοινοβουλίου ε, είναι σε πώς θα γίνει ο συντονισμός όλων αυτών, τι θα προχωρήσει πρώτο, τι θα προχωρήσει πιο πολύ κλπ. Γιατί, γιατί σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν και πολλά μπλοκαρίσματα. Ε, σε άλλους τομείς που υπάρχουν πολλά θέματα ε, δεν υπάρχουν τόσα μπλοκαρίσματα. Κύριε Μακοβέη, δεν είναι διαδικαστικό έτσι, δεν είναι. Ε, δεν θα είναι διαδικαστικό, το γνωρίζω. Εντάξει, τώρα είμαστε ειλικρινεί. Επί τη ουσία θέλω να μιλήσω. Όχι, δεν είναι διαδικαστικό αυτό, αφού μιλάτε, θέλετε να μιλήσετε επί τη ουσία, Μπορείτε να μου δώσετε 20 δευτερόλεπτα. Τι είναι, ψυχολογικό πόλεμο μου κάνετε τώρα. Αναφέρθηκε το όνομά μου, πρόεδρος. Γιατί δεν με βοηθάτε κι εσείς λίγο να προχωρήσουμε. Υπάρχουν εδώ εισηγητέ και όσοι συγητές που περιμένουν. Μερικοί έφυγαν βέβαια. Είναι άνθρωποι που δίνουν προτεραιότητα στα θέματα που συζητάμε, παρόλο που έχουν πολιτικά θέματα και στη χώρα τους και μας βοηθούν με υπομονή ε, και, ε, και συνεργάζονται με την Προεδρία και η Προεδρία κάνει ό,τι μπορεί. Σας παρακαλώ πολύ ας το αφήσουμε, ας το αφήσουμε εδώ. Ας λήξουμε τη συζήτηση αυτή με τους υπουργού σε αυτό το σημείο, εντάξει. Όχι. Ασφαλώς και δεν είναι εντάξει. Να πω το εξής και δεν θα μιλήσω για την ουσία. Εγώ υπερασπίζομαι τη χώρα μου και δεν δυσφημίζω κανέναν. Η κυρία Βουίλκστρομ είναι εδώ, η κυρία Γκρίσπεκ, όλοι όσοι ασχολούνται εντατικά με αυτά τα θέματα είναι εδώ. Γίνεται πολύ σκληρή δουλειά με την Προεδρία, να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι όμως οι φυσιολογικές και οι στιγμές αυτές, δεν είναι συνηθισμένες, όπως είπε ο Σκοέλιο. Η Προεδρία πάντως είναι σε επαφή με τους ηγητές, με τους κοιόδες. Παρακαλώ πολύ, επιμείνετε και μείνετε κινητοποιημένοι. Ευχαριστώ πολύ τους υπουργού, είναι η αρχή αυτή. Θα συνεργαστούμε στενά μαζί σας για την υπόλοιπη, κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης Προεδρίας σας. Ευχαριστώ πολύ. Και αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ψηφοφορία στις 11.45. Ευχαριστούμε τον κύριο Λένας για την ε, υπομονή. Διαλειτουργικότητα. Τριμερής διάλογος. Παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, ποιος είναι να αποχωρήσει, να αποχωρήσει ησύχως. Ναι, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε κύριος Μονομέλο. Θα είμαι... Κύριος Λένα, Θα είμαι σύντομος. Να κερδίσουμε λίγο χρόνο και από αυτό το θέμα. Ε, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Μέλο που είναι άρρωστος σήμερα και έτσι δεν μπορεί να έρθει. Μια σύντομη επικαιροποίηση λοιπόν των εξελίξεων στα θέματα της διαλειτουργικότητας από πλευράς μας. Έχει προχωρήσει το θέμα αυτό σημαντικά. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Λίμπε έγινε τον Οκτώβριο του 2018. Τέσσερις τριμερείς διάλογοι υπό την Αυστριακή Προεδρία με τελευταίο τον τριμερή στις 13 Δεκεμβρίου όπου καταλήξαμε σε μια καλή και ισορροπημένη συμφωνία ε, συμβαστική για τα εκκρεμή πολιτικά ζητήματα κοινό αποθετήριο ταυτότητας για την ταυτοποίηση και πρόσβαση για τις δυνάμεις επιβολής του νόμου ήταν σημεία συμφωνίας. Και για τα δύο αυτά λοιπόν έχουμε εξασφαλίσει τη διαφύλαξη της αποτελεσματικότητας του συστήματος αλλά και τον συσταλτικό ε, τη συσταλτική. Αν η κυρία Μακοβέ έχει την καλοσύνη να κάνει στο έξω από τη διάθεση της συναντήσης της σας ευχαριστώ. Διαφυλάξαμε λοιπόν την αποτελεσματικότητα του συστήματος αλλά και με συσταλτική χρήση των στοιχείων με τις απαραίτητες οικονομικές ασφαλιστικές δικλίδες που δεν θα επιτρέψουν την καταστρατήγηση των κανόνων σε σχέση με την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, σύστημα Schengen κτλ. Επίσης σημαντικό και ως κοινοβούλιο εμείς επιμείναμε σε αυτό, ήταν ότι ε, πείσαμε το Συμβούλιο να συμπεριλάβει μια ενημέρωση προς, τον, ε, προς το υποκείμενο των δεδομένων ότι έχει το δικαίωμα της ε, πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και της διόρθωσής τους. Κατόπιν αυτού σε κάποια σημεία που ακόμα δεν έχουν κλείσει συνεχίζει τη δουλειά σε τεχνικό επίπεδο, όπως το δικαίωμα προς ενημέρωση των υποκειμένων και θέση σε ισχύ των προτάσεων. Ε, χρειάζεται εδώ λίγο, λίγη πρόοδος, χρειάζεται υποστήριξη των θεσμικών οργάνων, τριμερής διάλογος και τελευταίο ελπίζουμε με τη Ρουμανία προβλέπεται στις 6 Φεβρουαρίου και πιστεύουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα αυτό. Αξιόλογο βέβαια το γεγονός ότι από το Δεκέμβριο του 2017 μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί όλη αυτή η πρόοδος που δεν θα ήταν δυνατή βέβαια χωρίς τη συνεργασία των σκιωδών και το είναι μεγάλη προσήλωση και σκληρή δουλειά του προσωπικού πολιτικών ομάδων, γραμματεία της ΛΥΜΠΕ αλλά και οργανώσεων όπως η ε, Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και λοιποί αποκεντρωμένοι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σου ευχαριστώ λοιπόν όλους και προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση των θεμάτων τον Φεβρουάριο για να ψηφιστεί τον Απρίλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λάνερτς. Κύριε Αβίξτρομ, θέλει το λόγο γι' αυτό ή κάτι άλλο. Σεσίλια, όχι γι' αυτό. Ακριβώς γι' αυτό και είναι πιστεύω η ώρα να το συζητήσουμε ως ομάδα. Νομίζω ότι υπό τον Χερούλτ ε, Λέναρς έχουμε προχωρήσει ως ομάδα πάρα πολύ και Ζερόμ οφείλω να σε συγχαρώ και να σε ευχαριστήσω για την πολύ ικανή αλλά και ευχάριστη καθοδήγηση που έδωσε στις εργασίες μας. Μαζί τα καταφέραμε και μαζί μπορέσαμε να φτάσουμε μέχρι τώρα στο σημείο που είμαστε στον τριμερή διαλόγο. Πολλέ από τι ε, ανησυχίε που είχαμε σχέση με τις αρχικές προτάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχική έκδοση του κειμένου, του κειμένου έχουν αντιμετωπιστεί με τρόπο ειλικρινή απλό, ιδιαίτερα όσον αφορά το κοινό αποθετήριο ταυτότητα στοιχείων ταυτότητα. Ιδιαίτερη δουλειά έχει γίνει επίση στη συμπερίληψη ασφαλιστικών δικλείδων για την ε, ορθή λειτουργία της διαλειτουργικότητας. Έκανε και ο εισηγητής όπως και όλοι μας ε, γενναιόδορες και ε, ειλικρινείς προσπάθειες για να ικανοποιηθούν τα μελήματα των άλλων και η ομάδα μου και εγώ ιδιαίτερο χαιρόμαστε για τη συμπερίληψη τροπολογιών για τα, την προστασία των παιδιών και την διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για πολίτες τρίτων χωρών ενημέρωση για την διακράτηση των στοιχείων ταυτότητας και δυνατότητα διόρθωση. Βεβαίως μένουν κάποια ζητήματα προς συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο. Προσβλέπω ωστόσο στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ελπίζομαι στη διάρκεια της θητείας, το δυνατό βέβαια προκειμένου να βελτιωθεί η κοινή χρήση στοιχείων ε, πληροφοριών που έχουν τα κράτη-μέλη σε θέση τους, αλλά και ταυτόχρονα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να διασφαλιστεί η ασφάλεια ε, και η αποτροπή κινδύνων για όλους μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ευχαριστώ και πάλι χαιρούν. Και ερωτώ, λέει ο Πρόεδρος, ε, αν θέλει κανείς τίποτα άλλο για τη διαλειτουργικότητα. Όχι, πολύ καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, χαιρούν. για όλη τη δουλειά και για την ενημέρωση. Προχωρώ. Σημείο 7. Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Εφαρμογή. Μια μελέτη ήταν αυτή. Περιμένω να έρθουν οι συνάδελφοι εδώ στο Προεδρείο για να κάνουμε και την παρουσίαση πρόκειται λοιπόν για κοινή συζήτηση για τη λειτουργία του κοινού συστήματος ασύλου. Απόφαση των συντονιστών να υπενθυμίσουν στην Επιτροπή την υποχρέωσή της για αναφορά δυνάμει των μέσων για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Η Επιτροπή λοιπόν καλείται να δώσει λεπτομερή επισκόπηση, την οποία βλέπετε και στα έγγραφά σας. Ο χρόνος μας μας πιέζει πολύ. Ας μην κάνω άλλη εισαγωγή λοιπόν εγώ. Και περνώ δίνοντας το λόγο αμέσω. Ψηφοφορίες είναι στι 11.45 έτσι. Ωραία. Ο κύριος Ράιν από την Επιτροπή. Κύριε Ράιν. Ναι, πιέζω λίγο. Γιατί οι ψηφοφορίε είναι σε 16.45. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν ε, κατάλαβα καλά, καλείται η Επιτροπή να παρουσιάσει μια σύντομη παρουσίαση ως προς τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στην υλοποίηση των ε, μέσων των νομοθετημάτων για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Πολύ ευχαρίστω. Και επίσης, επί τη ευκαιρία που προσφέρει αυτή η συζήτηση, θα ήθελα και να εξηγήσω γιατί κάποιες εκθέσεις εφαρμογής δεν έχουν υιοθετηθεί. Αυτό σύμφωνα με μια επιστολή που είχατε αποστείλει στον Επίτροπο Αβραμόπουλο. πριν τις δίκοπες των Χριστουγέννων. Η Επιτροπή βεβαίως ε, αντιμετωπίζει μεγάλη σοβαρότητα την υποχρέωση τη για ε, υλοποίηση και παρακολούθηση τη εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό ισχύει οπωσδήποτε και για όλα τα μέσα και νομοθετήματα τη συμφωνία για το κοινό σύστημα ασύλου και συνεχίζουμε το πράγμα αυτό παρά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσει ε, για την μεταρρύθμιση όλων των νομοθετημάτων του συστήματο ασύλου. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ άλλων οργάνωσε μια σειρά από συναντήσεις πραγματογνωμόνων των κρατών μελών για να συζητηθούν ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών, αλλά και ζητήματα σχετικά με την πρακτική υλοποίηση εφαρμογή των νομοθετημάτων. Ορισμένες περιπτώσεις γνώρισαν και την σύσταση επιτροπών κόντακ, όπως ονομάζονται, με συμπερίληψη και πραγματογνωμόνων και εμπλεκομένων φορέων και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλωστε και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής της Γραμματείας σας έχουν, ε, της Γραμματείας Επιτροπής σας έχουν προσκληθεί σε αυτές τις συναντήσεις. Μελέτες γίνονται για την εφαρμογή σε πρακτικούς όρους αλλά και σε νομοθετικούς την τη μεταφορά δηλαδή στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών στην οποία έχουν προβεί τα, τα κράτη-μέλη, έχουν γίνει αυτοψίες σε κράτη-μέλη με επισκέψεις που στόχο είχαν τη συζήτηση προβλημάτων στις εφαρμογές με τα κράτη-μέλη, με τους εμπλεκόμενους φορεί, εξέταση της κατάστασης αυτοψία ε, από πλευράς μας με στόχο ιδιαίτερα την, ε, τον εντοπισμό μέτρων που θα μπορούσαμε να λάβουμε για τη βελτίωση της κατάστασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό οδήγησε και σε αλλαγή των συστημάτων ή των πρακτικών των κρατών μελών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ε, η ΕΑΖΟ, το Γραφείο Υποστήριξης για το Άσυλο, έλαβε μέτρα εκείνο για να στηρίξει τα κράτη-μέλη. Σε λιγότερες ε, περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάστηκε να αναλάβει δράση αξιοποιώντα την νομοθεσία κατά των κρατών μελών σε περιπτώσει όπου σημειώνονταν σοβαρές παραβιάσεις τη νομοθεσία, δηλαδή όπου οι αλλαγές ήταν ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται να εφαρμοστούν. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθοδηγεί τις δραστηριότητες του Γραφείου Ασύλου σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της ε, στην υποστήριξη των κρατών μελών. Έχει στενή επικοινωνία και επαφή με το Γραφείο για το Άσυλο Έχουμε λειτουργική στήριξη προσφέρει στην Ελλάδα, επιχειρηματική στήριξη στην Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά και στην Κύπρο και σε άλλες χώρες. Ε, κατάρτιση στις αρχές των κρατών μελών, αλλά και καθοδήγησε πρακτικούς όρους στις αρχές διαχείρισης θεματών ασύλου. Δύο είναι τα πιο χτυπικά παραδείγματα η ανάπτυξη προδιαγραφών και δικτών υποδοχής όπως ονομάζονται στα κράτη-μέλη για την τήρηση κοινών προτύπων ε, σε πολύ λεπτομερείς και τεχνικού επίπεδου πολλές φορές ε, προδιαγραφές ε, για την υποδοχή αλλά και εκθέσεις για ενημέρωση και καθοδήγηση των κρατών ή κατευθυντήριες γραμμές που οδηγούν σε μια κοινή προσέγγιση για την αξιολόγηση της προστασίας. Και άρα σύγκληση και σε επίπεδο αναγνώρισης των ε, αιτήσεων ασύλου. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και προχωρά. Η διαδικασία παράβασης, επί παράβαση που έχει ξεκινήσει εις βάρος ορισμένων κρατών ως προς την εφαρμογή των κανόνων τώρα και θα ήθελα εδώ να αναφέρω κάποιες ε, στατιστικές σε γενικού όρου, 62 είναι οι ανοιχτέ υποθέσεις επί παραβάση των κρατών μελών για την νομοθεσία του ασύλου και αφορούν τη μεταφορά σε εθνικό ε, δίκαιο στην, ε, στα μεγαλύτερα ποσοστά τους. Είναι εκκρεμείς οι περισσότερες από αυτές. Μέχρι να τελειώσουν και οι μελέτες που ανέφερα νωρίτερα με την εξέταση των ε, μέσων ή των νομοθετημάτων εισαγωγής στο Εθνικό Δίκαιο των κρατών μελών. Επίσης, η αναφορά, η εκθέση περί αναφοράς. Οι διατάξεις περί αναφοράς που ανέφερα στην αρχή, που έχει ε, επικαλυστεί και η Επιτροπή σας, από την Επιτροπή την ε, υποβολή αναφοράς για την εφαρμογή του νομοθετήματος και πρόταση ή οδήποτε τροποποιήσεων θα χρειάζονταν. Κοιτάξτε, αυτό, μπορεί να συμβαίνει, αυτό που συμβαίνει και συμβαίνει πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσαμε ίσως να περιμένουμε μετά την υιοθέτηση ενός δεύτερης γενιάς κοινού συστήματος ασύλου ήταν ότι αναδείχθηκε μια προσφυγική κρίση η οτιδήποτε τροποποιησεων τονίζει τις ε, ιστερίες στα ελλείμματα στο κοινό σύστημα και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει πως θα χρειαστούν σημαντικές τροποποίησεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τις οποίες εκθέσαμε στην ανακοίνωση του Απριλίου του 2016 και οδήγησαν μάλιστα σε αρκετά φιλόδοξες τροπολογίες το Μάιο και τον Ιούλιο του 2016 στη συνέχεια. Ε, τροπολογίες οι οποίες ε, λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία που έχει συλλέξει η Επιτροπή. Ταυτόχρονα όμως ε, θεωρήθηκε πως θα διατάρασε αλλά και θα οδηγούσε σε σύγχυση της διαπραγματεύσεις που είναι εν εξελίξη, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τις νομοθετικές προτάσεις υιοθετούσε και τις τροποποιήσεις αυτών. Υπενθυμίζω ότι ο στόχος της έκθεσης ήταν ότι θέλαμε να εξηγήσουμε την ανάγκη νομοθετικών τροποποίησεων. Και προσθέτω ότι όλα τα ε, νομοθετήματα για το άσυλο συνοδεύονται από επεξηγηματικά υπομνήματα, όπως άλλωστε είχε ζητήσει και το Κοινοβούλιο, που εξηγούν αρκετά λεπτό μέρο τα προβλήματα που έχουμε συναντήσει στην υλοποίηση, στην εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο του κεκτημένου που έχουμε αυτή τη στιγμή και τους λόγους που μας οδηγούν στην τροποποίηση. Και μια και μας πιέζει ο χρόνος, θα σταματήσω εδώ. Ε, ευχαριστώ. Ελπίζω να μην ακούσατε τι ψιθύρισα. Δεν ήθελα να φανώ αγενής, αλλά όντως δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε και χρήσιμα. Ο δόκτωρ Φαν η δόκτωρ Φερνάντες ε, και η δόκτωρ... Ε, το έχετε πάρει το δακτορικό σας. Να λοιπόν, όλοι οι δόκτωρες εδώ, Ναβάρα. Η δόκτωρ Ναβάρα λοιπόν, EPRS, Milieu Limited και οι τρεις με ε, και οι τρει είναι συντάκτες της έκθεση «Το κόστος της μία Ευρώπη στην πολιτική ασύλου. Παρακαλώ. Ήδη στις 7 Ιανουαρίου παρουσιάσαμε μια πρώτη εκδοχή της μελέτης. Ε, σήμερα θα συνεχίσω από εκεί που είχα σταματήσει να σας πενθυμίσω ότι πρόκειται για το κόστος μη Ευρώπης που κοιτάει, εξετάζει ε, τα κενά και τα εμπόδια στη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ασύλο και το πώς όλα αυτά επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οικονομικούς παράγοντες και τα οικονομικά στοιχεία. Περνάμε στην επόμενη ε, διαφάνεια. Τα βασικά σημεία είναι ότι έχουμε εξετάσει τα κενά, όπως είπα, και τα εμπόδια ε, κατά τη διάρκεια όλου του ταξιδιού για άσυλο, ε, ξεκινώντας από την έλλειψη νομικό, νόμιμων ε, διόδων ε, και ελλείψεις στα, στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Δεύτερον, προφανές, αλλά πρέπει να το υπογραμμίσουμε, περισσότερη δράση ε, στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των κρατών ε, μελών ε, και σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τρίτον, για να επιτύχει αυτό χρειαζόμαστε ευρύτερη δράση στον τομέα του κράτους δικαίου, τον έλεγχο των συνόρων, την νόμιμη μετανάστευση και την εξωτερική πολιτική. Όπως είπαμε, η μελέτη αυτή δεν σχετίζεται άμεσα με τους νομοθετικούς φακέλους που συζητώνται αυτή τη στιγμή. Εξετάσαμε όλο το, όλη τη διαδρομή του ασύλου. Το βλέπετε εδώ. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Τα κενά και τα εμπόδια που, που εντοπίσαμε είναι παρόμοια αυτά που βλέπετε εσείς εδώ. Έλλειψη νόμιμων μορφών εισόδου, έλλειψη βιώσιμης κατανομής επιμερισμού της ευθύνης, ανεπαρκείς συνθήκες ε, ε, εισδοχής, ε, αδύναμη εφαρμογή των διαδικασιών, περιορισμένες υπηρεσίες ε, για την διευκόλυνση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, περιορισμένη στην εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής και απουσία μηχανισμών παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες στις οποίες επιστρέφονται και γενικότερα μη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα τα δούμε αργότερα. Το βλέπουμε εδώ. Ε, κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στις επιπτώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ατομικό επίπεδο ε, και ε, τις επιπτώσεις σε οικονομικό επίπεδο για τα κράτη-μέλη. Όπως δείτε, βλέπετε εδώ τα, τα τρία αυτά βέλη κατά τη διάρκεια της όλης διαδρομής. Ε, ε, καταρχήν πρώτης αύξηση υπάρχουν θέματα α, ε, απουσίας ε, νομιμών διόδων, Γι' αυτό οδήγησε σε 8.000 άτομα θα να χάσουν τη ζωή τους το 2016-2017 και παρόμοιο αριθμό το 2018 υπάρχει περιορισμός ε, στην, ε, ε, στην άσκηση του δικαιώματος στο άσυλο λόγω των επιστροφών εν θερμό κλπ. Το δικαίωμα του ασύλου επίσης υποσκάπτεται εξαιτίας ευαδυναμιών στο σύστημα του Δουβλίνου και διαφορές ανάμεσα στις διαδικασίες μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης υπάρχουν και τα δικαιώματα των παιδιών που δεν τη χάνουν σεβασμού. Όταν γίνεται η αναγνώριση από την άλλη μεριά, υπάρχουν ένας, υπάρχει ένα ορμό οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, μεταξύ αυτών το δικαίωμα στην εργασία, που δεν ε, υλοποιούνται εξαιτία του ότι δεν υπάρχει παρκή στήριξη σε αυτού του τομεί. Επίσης, ενεχόμενες άδικες ε, διαδικασίες, ε, αποφάσεις επιστροφής μπορούν επίση να υποσκάψουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μαζί με όλα αυτά, αυτές τις προσβολές στα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις σε επίπεδο των κρατών μελών. Βλέπετε εδώ ε, τον πίνακα αυτό, να τα διατρέξουμε. Ορισμένα εμπόδια και δυναμίες αυξάνει τον, τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση παρατυπίας αυξάνουν τα κόστη σε ό,τι αφορά το, τον έλεγχο ε, της παραμετανάστευσης και του εμπορίου ανθρώπων. Ε, δεύτερον, έχουμε θέματα κατανομής ευθύνη, κόστη ε, εξαιτία της ε, του, του φορολογικών εσόδων. Τέταρτον, συνθήκες ζωής και διαβίωσης, ε, κακής ποιότητας, ε, μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας κλπ. Πέμπτον, ε, κόστος εξαιτία των ετοιμάτων, ασύλου, επιστροφών κλπ. Τρια, περίπου 49 δισεκατομμύρια το χρόνο στο συνολικό κόστος. Ωραία. Πολιτικές επιλογές τις γνωρίζετε σε μεγάλο βαθμό, πολλοί από εσά. Πρώτον, η θέσπιση ανθρωπιστικών θεωρήσεων, όπως έχετε προτείνει και εσείς, το σκέφτεται η Κομισιόν. Διεύρυνση της εντολής του Ευρωπαϊκού, Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης του Ασύλου. Τρίτον, σημαντική δυνατότητα, διότι αυτή τη στιγμή, ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν ήμασταν έτοιμοι πρέπει να εφαρμόσουμε και να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία του κοινού συστήματος ασύλου. Τέταρτον, οι ατομικές επιλογές και προτιμήσεις να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη όταν εντοπίζεται το κράτος που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία του αιτήματος ασύλου. Πέμπτον, να ενθαρρύνουμε πρόσβαση στην ε, ένταξη και την ε, εργασία. Έκτον, να διασφαλίσουμε ότι κάποιο θα λογοδοτεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για του οικονομικού παράγοντε. Περαιτέρω δράση προ αυτές τις κατεύθυνσει θα διασφάλιζε καλύτερη συμμόρφωση με τα διεθνή δικαιώματα και αξίε. θα στήριζε τι τρίτε ε, χώρε, ε, θα μείωνε τα ποσοστά παράνομη μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μείωνε το κόστος της ασφάλειας των συνόρων, θα βελτίωνε τη διαχείριση, την αποτελεσματικότητα και το συντονισμό των διαδικασιών ασύλου, θα βελτίωνε την οικονομική και κοινωνική ένταξη των ετούντων και των προσφύγων, ε, θα δημιουργούσε περισσότερη ε, εργασία και θα ενίσχυε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επόμενη διαφάνεια. Τώρα όλα αυτά βέβαια ως δράσεις θα έχουν και κόστος, ε, ανθρώπινο και οικονομικό κόστος, γιατί θα χρειαζόταν για να βελτιωθεί η ικανότητα της υπηρεσίας, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου και των Εθνικών Αρχών Ασύλου, ε, προκειμένου να εντάσσονται καλύτερο, καλύτερα οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Ε, θα χρειαζόταν από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρακολουθηθούν και να αξιολογηθούν οι συμφωνίες επανεισδοχής, θα έπρεπε να ενισχυθούν τα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών και να ε, δημιουργηθούν καλύτερα προγράμματα ένταξη, για παράδειγμα, γλωσσική εκμάθησης. Το συνολικό κέρδος που θα προέκυπτε από αυτές τις ε, πολιτικές θα ήταν περίπου 22,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατ' έτος. Λαμβάνοντας υπόψη και τα κόστη βέβαια αυτών των πολιτικών. Δεν έχουμε αξιολογήσει όλες τις πολιτικές δυνατότητες, τις πολιτικές επιλογές που έχουμε, αλλά ε, θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου για την... Ε, αν, θε, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις μπορούμε να απαντήσουμε και εγώ και ο συναδελφός μου. Ε, Θα στηριχθώ στην... Ε, θα παρουσιάσω μια οικονομική αξιολόγηση που έχει κάνει η μελέτη μας για να σας δώσω και τα οικονομικά στοιχεία πίσω από τα λόγια των συναδέλφων σήμερα. Η μελέτη λοιπόν αυτή είναι μοναδική φιλόδοξη. Κοιτάει την περίοδο πριν από την άφηξη έως μετά την υποβολή της ε, αίτησης. Κοιτάει που υπάρχουν ζητήματα, νομοθεσία, ε, οδηγία, νομικά ζητήματα, οικονομικές συνιστώσεις όπως και νομικές Πληροφορίες παίρνουμε από τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές Ασύλου αλλά και από άλλες πηγές πολύ ενδιαφέρουσες που έχουμε ενσωματώσει. Στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης και λοιπόν με τα οποία έχουμε κατασκευάσει βάση δεδομένων με διάφορους δείκτες πάνω στους οποίους στηρίξαμε τις εκτιμήσεις και προχωρώ παράλληλα με την ε, κατασκευή αυτή της βάσης δεδομένων ορίσαμε ένα πλαίσιο. Είπαμε ότι θέλουμε να εστιαστούμε, αποφασίσαμε να εστιαστούμε σε εννέα κενά και ελλείψεις που εντοπίζουμε ως κύρια, γιατί δεν είναι τα μοναδικά, κενά ή φραγμοί που οδηγούν σε συγκεκριμένα ζητήματα με βάση τα οποία μπορούμε να εκτιμήσουμε την όλη προβληματική. Έτσι λοιπόν, Έχουμε κακή διαχείριση και συντονισμό πρώτον. Δεύτερον, ε, κακό, κακή καταγραφή των αναγκών και προτιμήσεων. Μικρή προξ, προβλεψιμότητα τρίτον, μια ιδέα που προέρχεται από μια μελέτη του ΟΣΑ που εξετάζει την αποτελεσματικότητα των ε, διαδικασιών, ε, των δικαστικών διαδικασιών και της προβλεψιμότητας, δηλαδή τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα κράτη-μέλη που οδηγεί σε χαμηλή προβλεψιμότητα και άρα αναποτελεσματικότητα. Και βέβαια ζητήματα ξενοφοβίας και ρατσισμού που πάλι προερχόνται από άλλη μελέτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έξι κατηγορίες συνεπειών έχουμε καταγράψει. Υπάρχουν και άλλες βέβαια που δεν καταγράφονται στην οικονομική αξιολόγηση, όμως έχουν αντανάκλαση στην κοινωνία και την οικονομία, αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Και αυτό το βλέπετε εδώ σε αυτούς τους ε, πίνακες. Και προχωρώντας στην επόμενη διαφάνεια, εδώ βλέπετε τα εννέα κενά και οι φραγμοί πώς αντιστοιχούν στις κατηγορίες συνοποιών και τα αποτελέσματα συνολικά. Για παράδειγμα, όταν δεν υπάρχουν ένδικα μέσα ή βοηθήματα, βλέπετε ότι αυτό έχει συνέπειες σε κάθε μία από τις έξι κατηγορίες συνεπειών. Με τη χαρτογράφηση αυτή έχουμε κάνει και τις δικές μας εκτιμήσεις στη συνέχεια. Και έτσι θα σας ε, δώσω, αν έχω το χρόνο, τις επιλογές πολιτικής Επτά διαφορετικές επιλογές πολιτικής έχουμε αξιολογήσει εμείς, εκτιμήσει. Ανθρωπιστική βίζα. Με, ευρωπαϊκή, με αξιολόγηση ευρωπαϊκής ε, προσθέμενης αξίας, όπως έχει προτείνει η ΛΥΜΠΕ. Και εξηγούμε εδώ το κόστος που βλέπουμε να συνδέεται με τις επιλογές. Καταρχάς, ανθρώπινοι πόροι που χρειάζονται για την εξέταση και επεξεργασία της αίτησης και τα λοιπά ε, Νομική υποστήριξη, διερμηνία, εξέταση και στα ωφέλη βλέπουμε ε, έχουμε θέσει ως υπόθεση πως μειώνεται κατά 20% το κόστος που θεωρούμε δεδομένο με βάση το status quo. Με αυτό σημειώνουμε βελτίωση κέρδος, δηλαδή κατά 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για την ε, Ευρώπη συνολικά σε σχέση με το να μην υπήρχε αυτή η επιλογή. Και καθώς δεν έχω χρόνο προχωρώ στην τελευταία διαφάνεια, τα συμπεράσματα. Εδώ όπου βλέπουμε συνολικά ότι τα κενά και οι φραγμοί στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου αντιστοιχούν σε σημαντικό κόστος για το ε, νηδιώτη αλλά και την κοινωνία. Αρνητικά ευρήματα υπάρχουν, αλλά στα θετικά μπορούμε να επισημάνουμε πως επιλογές με πολιτικές ε, παρεμβάσεις έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί έτσι να καλύψει τα κενά αυτά, να αποκομίσει ωφέλη. Είναι πολύ σημαντικό να ε, εξεταστούν κριτικά αυτές οι επιλογές. Ε, χρειάζεται περαιτέρω μελέτη βέβαια και ανάλυση και ε, για να είναι αποτελεσματικές αυτές οι επιλογές πρέπει να επιλεγούν εκείνες οι οποίες δίνουν απαντήσεις στους λόγους για τους οποίους έχουν συνέπειε τα κενά και οι ελλείψεις και οι φραγμοί. Δηλαδή πρέπει να βελτιωθεί η προβλεψιμότητα της διαδικασίας του ασύλου, να ενισχυθεί το δικαίωμα για εργασία και να μην υπάρχουν διακρίσεις Ευχαριστώ πολύ και ο Στίβεν Ράιεν θα μας μιλήσει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να απαντήσει και στα δεδομένα του, της κυρίας Ναβάρα ε, και της δόκτωρος Μένα Φερνάντες. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ακολουθήσαμε συνοπτικές διαδικασίες, ε, θα πρέπει να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Άλλοι, πάμε. Δύο μέλη ζητούν το λόγο, Γκρίσπα και Λόπες Αγγιλάρη. Η Νάταλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ εντάχει, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή την ε, παρουσίαση, αν και δεν είχαμε χρόνο να συζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς έχει η κατάσταση στην Ευρώπη και να δούμε το κόστος της μη Ευρώπης στις ε, διάφορες συνεδριάσεις όπως βλέπουμε με τα fake news και τις ε, διάφορες απειλές των ε, εθνικιστών. Τα στοιχεία ε, είναι εύγλωτα σε σχέση με το στάτους κουβό, σε σχέση με το άσυλο, 50 δις ευρώ. Το λέμε σε όλες τις συνεδριάσεις, θέλουμε να προχωρήσουμε στην αναθεώρηση του δικαιώματος χορήγησης ασύλου, αλλά δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε ότι τα πράγματα δεν έχουν μπλοκαριστεί από το Κοινοβούλιο, αλλά από το Συμβούλιο. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, στο πρώτο τμήμα της έκθεσης μιλάτε για την έλλειψη νομικών οδών και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι άνθρωποι σε σχέση με τα ευεργετήματα των διακινητών. Θα μπορούσατε να μας ε, αναλύσετε εντάχει και γραπτός ως προς την ε, εκτίμηση για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις μπορεί να επιλύσει εν, μέρος, ε, ε, ε, εν μέρη συγγνώμη, το ζήτημα και αν ναι πώς. Σας ευχαριστώ πολύ Νάταλη. Εντάχει ο, ο κύριος Αγγιλάρ, ναι, γνωρίζουμε ότι είμαστε πολύ περιορισμένοι από χρόνο. Αλλά θα ήθελα να αποτανθώ στους εκπροσώπους της Επιτροπής ακούσαμε για διαδικασίες επί παραβάση. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτό το χάσμα μεταξύ του νομικού πλαισίου και της συμπεριφοράς των κρατών μελών. Αυτό δείχνει περιφρόνηση, άμεση περιφρόνηση αλλά και παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου που έχει τεθεί σε εφαρμογή και είναι δεσμευτικό αυτό το πλαίσιο. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες για τις διαδικασίες επί παραβάση. Είναι δημοσιοποιημένες. Υπάρχει κάποιο κράτος μέλος που δεν υπόκειται σε αυτή τη διαδικασία για παραβίαση του Ευρωπαϊκού Πακέτου για το Άσυλο. Είδαμε και αυτή την παρουσίαση για την κατάσταση και μία από τις προκλήσεις, ένα από τα ζητήματα, είναι ότι οι επιστροφές δεν είναι αποτελεσματικές. Αυτό αναφέρθηκε. Σπάνια αναφέρεται ότι ο αριθμός των επιστροφών είναι εντυπωσιακός. Σε πολλές χώρες υπάρχουν περισσότερες επιστροφές παρά παράνομοι μετανάστες που τα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι εκεί. Πόσο σημαντικός είναι ο αριθμός ως προς τις πραγματικές επιστροφές, γιατί πολλές φορές ε, είναι εντυπωσιακό ο αριθμός. Η ε, Νάταλη και Χουάν υπέβαλαν τις ερωτήσεις. Ε, είναι πολύ σημαντικές ψηφοφορίες και θα πρέπει να απαντήσετε γραπτώς. Η μία ερώτηση απευθύνεται άμεσα στην Κομισιόν, αλλά δεν γίνεται να απαντήσετε προφορικά. Μπορείτε να απαντήσετε γραπτός, θα σας δώσουμε τα email Ευχαριστούμε τον Στίβεν και την ομάδα και τους δύο βουλευτές που υπέβαλαν ερωτήσεις. Αρχίζουμε τις ψηφοφορίες σε ένα λεπτό. Είναι πολύ ευαίσθητα τα θέματα. Θα ήθελα να έχετε τις κάρτες σας. Αν δεν τις έχετε, πηγαίνετε να τις πάρετε. Ή να μου το πείτε, εν πάση περιπτώσει, αν δεν τις έχετε. Thank you. And we'll start in, uh, a few seconds. Σε μερικά δευτερόλεπτα ξεκινάμε. Colleagues, everyone ready? We can... Uh, Μπορούμε να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Κάνουμε μια μικρή επαλήθευση πρώτα για να ξεκινήσουμε. Yeah, okay. Okay, colleagues, um, we begin on the, the voting. Uh, With Ξεκινώ λοιπόν με το σημείο 9, αγαπητοί συνάδελφοι. Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Αξιωματικών Συνδέσμων Μετανάστευση Αναδιατύπωση, κυρία Κέντζε. Θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, Κλοντ, ευχαριστώ πολύ, γιατί ήθελα μόνο σύντομα να ευχαριστήσω τη γραμματεία και όλο μας το προσωπικό για το πνεύμα συνεργασίας και την διαθεσιμότητα που επέδειξαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Σεσίλ και πάμε ψηφοφορία λοιπόν. 39 αρχίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Παρακαλώ όλοι να πατήσετε σας και να αρχίσετε τη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τις κάρτες σας τις έχετε. Πέρας. Απερίφθη 40. Αρχίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική πρώτη. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 2. Αρχίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 3. Αρχίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 125. Αρχίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. 4. Συμβαστική 4. Πέρας. Εγκρίνεται 127. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 5. Αρχίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 128 ως προσθήκη, παρακαλώ. Πέρας. Απερίφθη. 147 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 150. Πέρας. Απερίφθη, συμβαστική 6, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Αρχίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 160. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 8. Ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται συμβαστική 9 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται 29 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται 163 ψηφίζουμε πέρας Απερίφθη. 173 ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη 174 ψηφίζουμε. Πέρας. Δέκα συμβαστικοί ψηφίζουμε. Πέρας. Συμβιβαστική 11. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 180. Ψηφίζουμε. Το ΕΛΚ έχει έναν υπεράριθμο σε αυτήν. Δεν χρειάζεται να σε συλλήφια, όποιος και να είναι. Να βγάλει την κάρτα του. Τώρα σας λείπει ένας. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Ψηφίζουμε. Πέρασε εγκρίνεται. 190 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απερίφθη συμβαστική 13 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται 197 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απερίφθη. Να πάμε on block μέχρι την 201. 198 μέχρι 201 παρακαλώ. όμως, Όχι. Όχι. 198. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. 199 ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. 200 ψηφίζουμε. Πέρας. 201. ψηφίζουμε. Πέρασε. Απερίφθη. Τροπολογία 14, συμβαστική, ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 15 συμβαστική ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 204 ψηφίζουμε. Πέρας. Απεριφθεί. λογική 41. πέρας απεριφθεί 42 πέρας Απερίφθη 50, 46 ψηφίζουμε πέρας απεριφθεί συμβαστική 16 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται τροπολογία 51 ψηφίζουμε πέρας απερίφθη 17 συμβεβαστική 17 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται συμβεβαστική 18 πέρας Εγκρίνεται συμβαστική 19. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 20 συμβαστική 20. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 21. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 22. 22 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 23 συμβαστική. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 24. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 71. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 73 και 8. Ψηφίζουμε μαζί. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβαστική 25. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 76. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη 77. Πέρας. Απερίφθη 26. Όχι, την 78 πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη 26 συμβαστική. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 82. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απεριφθεί 81 παρακαλώ. Πέρας. Απεριφθεί συμβαστική 27. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται συμβαστική 28. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 29. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται τροπολογία 19. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη συμβαστική 30. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 31. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 32 συμβαστική. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 33. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 34 συμβαστική. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 34 συμβαστική. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται και αυτή. Το σύνολο του κειμένου πώς τροποποιήθηκε, ονομαστικά παρακαλώ. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. 38 υπέρ, 11 κατά, 5 αποχές εγκρίνεται και έτσι Και τώρα η εντολή για την άρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρας. 39 υπέρ, 13 κατά. Δύο εποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο ε, προσψήφιση σημείο. Θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, μη πηβήτα 3. Συγγήτρια κυρία Βαλέρο. Μποντιλ, θέλεις το λόγο? Όχι. Περνάμε κατευθείαν στις ψηφοφορίες. Συμβιβαστική υπαριθμόν 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90. άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Τροπολογία υπαριθμών 90. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Ναι, ναι, 90. Ψήφισαν όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9, υπέρ. Συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 91. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 92. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 93. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 94. Άρχεται. Λίγη. Απορρίπτεται. 95. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. 96. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. 97. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ομαδικά τις 98 ως και 103. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγοι, Απορρίπτεται, απορρίπτονται. Συμβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 121. Τροπολογία 121. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 13. Άρχιτη ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3. Λήξη της πληροφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 127. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Ταυτόσημες οι 128 και 129 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγοι απορρίπτονται. Εκτιμώντας 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγοι απορρίπτεται. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγοι. Εγκρίνεται 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. 19 άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 21. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται 22 άρχεται. Λίγη. Απορρίπτεται 23 άρχεται η ψηφορία. Λίγη. Απορρίπτεται 24. Λίγη. Εγκρίνεται. 26 άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 27 άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 28 άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 29. Έναρξη ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Πόσα, πόσες παραγράφους έχουμε στην, στην αιτιολογική έκθεση, πολλές. 30. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 31. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 33. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 34. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 35. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 36. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 1. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 40. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 41. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 42. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 2. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 44. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 45 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 46 έναρξη. Λήξη. Κρατήστε το χέρι σας στη συσκευή. Μην το αποσύρετε. 47 έναρξη. 46 εγκρίθηκε. 46 εγκρίθηκε. 47 τα Έναρξη. Λίγη. Λήξη. Απορρίπτεται. 48. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Ψήφισαμε λάθος εκεί. 49. Ε. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 50. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 3. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 51. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται 52. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 53. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 54. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 55. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 56. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 57. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 58. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 59 έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 60 έναρξη. Λήξη. Δεν ξέρω γιατί με κινηματογραφούν, με καταγράφουν στην κάμερα. Τόσο ενδιαφέρον είναι αυτό που κάνουμε. 61 έναρξη. Λήξη. εγκρίνεται 62 έναρξη λήξη εγκρίνεται 63 έναρξη λήξη απορρίπτεται 64 έναρξη λήξη εγκρίνεται 65 έναρξη λήξη Απορρίπτεται. 66 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 67 έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 4 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 68 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο στο σύνολό του. Έναρξη. Με ονομαστική ψηφοφορία. Λήξη. 38 ψήφοι υπέρ, 4 κατά 10 αποχές εγκρίνεται το κείμενο. Συγχαρητήρια στον, στην εισηγήτρια. Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και τη κοινή δήλωση που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και επί των αποκεντρωμένων οργανισμών. Επόμενο θέμα. Η συγγήτρια κυρία Γραπίνη. Θέλετε το λόγο. No. Okay, thank you. So, we go to... Ωραία. Προπολογία, 2 και 6 μαζί, unblock, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται. Ένα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 3 άρχεται. Πέρας εγκρίνεται 4 άρχεται πέρας εγκρίνεται 5 άρχεται λήξη εγκρίνεται 7 άρχεται πέρας απορρίπτεται 8 άρχεται Πέρας. Εγκρίνεται. 9. Ναι, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 10. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 11 υπέρ, ε, συγγνώμη, άρχεται, πέρας εγκρίνεται 12 άρχεται πέρας εγκρίνεται 13 άρχεται πέρας εγκρίνεται 14 άρχεται πέρας εγκρίνεται 15 άρχεται Πέρας. Και εγκρίνεται τελική ψηφοφορία με ονομαστική, η οποία και αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 54 υπέρ, κανείς κατά, καθόλου αποχές. Να συγχαρούμε την εισηγήτρια. Το επόμενο είναι μία ψηφοφορία για το κεντρικό σύστημα για πληροφορίες ποινικού δικαίου για, υπο, για υπηκό συγγνώμη τρίτων χωρών και απάτριδες. Ο Ντάνιελ Ντάλτον είναι ο εισηγητής και πριν ε, προχωρήσουμε ο κύριος Ντάλτον θέλει το λόγο. Εντάχει θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν πολύ σκληρά. Δύο χρόνια πριν, όταν ανέλαβα αυτό το θέμα, θεώρησα ότι θα ήταν κάτι το εύκολο, αλλά ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες κάνανε συμβιβασμούς και πιστεύω ότι θα περάσει σήμερα με βάση και τους συμβασμούς που έκαναν όλοι, που ήταν δύσκολοι για τους πάντες. Τίποτα δεν είναι εύκολο στη Λίμπε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και έπονται και άλλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε απευθείας στην ψηφοφορία όπως ε, αποφασίστηκε. Άρχεται η ψηφοφορία για ολόκληρο το κείμενο. What's that All right, two. Sorry. My apologies. Ναι, ζητώ συγγνώμη, δύο είναι οι ψηφοφορίες, διορθώνει ο πρόεδρος. Πέρας καταρχήν. Εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ 11 κατά και 9 αποχές. Και τώρα ψηφίζουμε την οδηγία. Σας ζητώ συγγνώμη, συγγνώμη προς τον εισηγητή δικό μου το λάθος. Τώρα ψηφίζουμε για την οδηγία. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την οδηγία ψηφίζουμε τώρα. Άρχεται. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται 37 υπέρ 8 κατά και 9 αποχές. Να συγχαρούμε τον εισηγητή time. Λήξη της ψηφοφορίας. Αρχίζουμε στις 4. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. <laughs> You just...